Hello, dear colleagues. We are going to start the meeting. Hello. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Abbiamo concluso stamattina. Κάτι ολοκληρώσαμε σήμερα στο τέλος τη συνάντηση των συντονιστών και εξετάσαμε τα σημεία που περιλαμβανόταν στη ημερήσια διάταξη. Θα σας πω ποιες είναι οι αποφάσεις των συντονιστών για τη διαδικασία, για την ενασχόληση από το Κοινοβούλιο και με τα φορείς ε, που είναι questional submissions όπως τα λέμε στα αγγλικά. Ακριβώς ε, υιοθετήσαμε την διαδικασία μέσω των συντονιστών και που διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη με τη συνεργασία της Γραμματείας. Στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής ε, τα στοιχεία αυτά θα μπουν σε ένα κατάλογο και θα ψηφίσουν τα μέλη της Επιτροπής. Και έτσι να απαντήσουμε σε όσα λέει η νομική υπηρεσία που με έκανε παρατηρήσεις για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε περίπου για ένα εξάμηνο. Όσον αφορά τώρα τις δύο αναφορές Πρώτα την αναφορά 0301 του 2011 για την ε, καταστροφή στο Σμόλενσκ. Τι αποφάσισαν οι συντονιστές. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ε, από νομική υπηρεσία και από την απάντηση της Επιτροπής να προτείνουν ότι πρέπει να κλείσει αυτό και θα μπει στο παράτημα 2 ακριβώς ε, της Επιτροπής μας και διακόπτει η Πρόεδρος. Κολέγα, Ζητάει το λόγο ο συνάδελφος στο σημείο αυτό. Uh, uh ευχαριστώ. Θέλω να θίξω τρία σημεία. Πρώτον, για την αναφορά για το Σμόλενσκ. να υπενθυμίσω ότι η νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν ήταν αρνητική και η αναφορά σε συνάντηση των συντονιστών θεωρήθηκε παραδεκτή. Δεύτερον, ούτε ο κύριος Τσίτσεστερ ούτε εγώ μπορούσαμε να παρευρεθούμε σήμερα το πρωί στην συνεδρίαση των συντονιστών. Ζητήσαμε να αναβληθεί λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η παράκλησή μας απορρίφθηκε. Το βρίσκω κάπως ε, ε, περίεργο αυτό, απαράδεκτο θα έλεγα. γιατί θα θέλαμε να μπορέσουμε να επιχειρηματολογήσουμε. Φυσιολογική διαδικασία είναι όταν υποβάλλεται έτοιμα για αναβολή λόγω απουσίας. Το αίτημα αυτό γίνεται αποδεκτό. Τώρα δεν έγινε αποδεκτό και λυπάμαι γι' αυτό. Και το τρίτο είναι το ότι σας υπενθυμίζω ότι η αναφορά πρώτον θεωρείται παραδεκτή, δεύτερον υπεγράφει από μισό εκατομμύριο άτομα στη χώρα μου και πέραν της χώρας μου. Ίσως και περισσότεροι να την έχουν υπογράψει. Ποτέ στο παρελθόν έχει υπάρξει μια αναφορά που να θεωρείται παραδεκτή με τόσο βάρος και, κατόπιν να κλείνει χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στους αναφέροντες να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τη γνώμη τους. Αυτό είναι σχεδόν σκάνδαλο. Και καλό τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής μας και εσάς κυρία Πρόεδρε να απορρίψετε την ε, πρόταση των συντονιστών οι αναφέροντες ε, τουλάχιστον πρέπει να ακουστούν. Δεν προκαταλαμβάνω το αποτέλεσμα της συζήτησης. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε την άποψη των αναφερόντων. Όχι να ακούσουμε τις απόψεις των κυβερνήσεων ή διαφόρων ισχυρών συμφερόντων. Θα καλούσα λοιπόν τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής μας να απορρίψουν την πρόταση των συντονιστών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Στάσφος Γιάρ θα λάβει το λόγο, αλλά να σας πω ότι η απόφαση των συντονιστών που βασίστηκε σε τρεις ε, συλλογισμούς. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή γνωμοδότησε αντίθετα όσον αφορά την αρμοδιότητα των ε, θεσμικών οργάνων. Εδώ λοιπόν έδειξε επίσης ότι αυτή τη στιγμή τρέχει μία, διαδικ... μία νομική διαδικασία, δικαστική μάλλον και εμείς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε δεν εξετάζουμε τις αναφορές. Περιμένουμε την εκδίκαση. Και το τρίτο είναι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που εκφράζει την αντίθεσή της σχετικά με την αρμοδιότητα της Ένωσης. Οι τρεις λόγοι λοιπόν είναι αυτοί. Στο παράτημα Β, στις παραδεκτές ε, την ε, συμπεριλάβαμε, δεν επανασυζητήσαμε αν είναι παραδεκτή όχι, αλλά γιατί μπαίνει στο παράρτημα Β. Μετά από τις απαντήσεις που λάβαμε και που μόλις ανέφερα, ε, ε θεωρείται ότι έκλεισε αυτή η αναφορά. Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφο Γιάρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για το περιεχόμενο δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Πολύ σωστά περιγράφει το θέμα. Δύο-τρεις ε, επισημάνσεις και ίσως ε, διορθώσεις. Δεν είναι πρώτη φορά που μας απασχολεί. Μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα αυτή η αναφορά. Έχουμε τη γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας έχουμε την απάντηση, την απάντηση της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά τα αποτιμήσαμε και η πλειονότητα των ε, συντονιστών αποφάσισε να κλείσει την αναφορά. Ίσως να δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το κάναμε αυτό κάποια στιγμή που έλειπε μια πολιτική ομάδα. Δεν ισχύει αυτό. Το θέμα αυτό είχε αναγγελθεί στην ημερήσια διάταξη. Αν ε, θα ήθελα να είμαι προέρετος, θα μπορούσα να πω ότι ορισμένοι ε, κάνουν πολιτική της ε, καινής θέσης. Δηλαδή λείπουν για να μην μπορέσει να συζητηθεί το θέμα. Και ανεξάρτητα από τι συμφωνήθηκε στους συντονιστές, η Επιτροπή έχει δυνατότητα να επικυρώσει ή να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση. Και τελευταίο κάθε αναφορά που μας υποβάλλεται και που αποφασίζουμε να κλείσει, υπάρχει δυνατότητα, αν προκύπτουν νέα στοιχεία, να την ξανανοίξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να αντιτεθώ στην εντύπωση που δημιουργείται, που επιχειρείται να δημιουργηθεί, δεν είναι καμία προσπάθεια πολιτικού ελιγμού, είναι επί της ουσίας απόφαση. Χρειαστήκαμε μήνες για να φτάσουμε σε αυτήν την κατάληξη και η κατάληξη είναι η σωστή και αρμόζουσα κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Όκεν. Δύο διορθώσεις. Δεν συμφωνήσαμε γι' αυτό. Εγώ ήθελα να μείνει ανοιχτή η αναφορά και πίστευα πως θα ήταν ευγενές κάτι τέτοιο, ευγενικό. Δεν ε, απέρριψαν το έτοιμά σας όλοι. Και δεύτερον, δεν είναι σωστό ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα ανεκρεμή ενώπιον των δικαστηρίων. Έτσι έχει η κατάσταση με τον ε, διαμεσολαβητή. Εμείς μπορούμε. Μόνο ο Ombudsman δεν μπορεί να ασχοληθεί με κάτι που εκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και τα αντίστοιχα άρθρα που μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε μια τέτοια υπόθεση. Ευχαριστώ τους αδελφούς. Λιγκούτκο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Με μικρόφωνο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δεν έχει το μικρόφωνο του ο μιλητής. Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε περάσει πολύ χρόνο συζητώντας ε, το θέμα αυτό. Πολύ λίγο χρόνο δαπανίσαμε. Ε, μας κόψατε όταν θελήσαμε να αναπτύξουμε το θέμα. Και επίσης, η νομική πραγματογνωμοσύνη του Κοινοβουλίου απεφάνθη ε, όχι αρνητικά. Ήταν θετική η, απο, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Προτιμώ η απόφαση να ληφθεί από την ε, Επιτροπή στο σύνολό της και όχι μονάχα από δύο-τρεις συντονιστές. Πρόεδρος. Νομίζω πάντως ότι η Επιτροπή είναι αυτή που έχει πάντα το, την τελευταία λέξη και ε, ε, εάν οι συντονιστές δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους και δεν έχουν κοινή θέση, τότε οπωσδήποτε το ζήτημα παραπέμπεται στο σύνολο της Επιτροπής. Εγώ ε, θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή εάν είναι υπέρ της προτάσεως ή κατά της προτάσεως των συντονιστών. Ποιος είναι υπέρ του να κλείσει το θέμα αυτής της αναφοράς για το Σμόλενσκ. Πώς... Και κοντράριο. Κατά. Να μην κλείσει. Τόδηση βότη. Δώδεκα. Έχουμε λοιπόν 12 ψήφου ψήφους υπέρ, 4 ψήφους ε, κατά και μία αποχή. Επομένως, επιβεβαιώθηκε η απόφαση έτσι όπως είχε εξαγγελθεί στην αρχή ε, της ε, συνεδριάσεως. Περνάμε επομένως στο σημείο 3 των συντονιστών. Οι συντονιστές λοιπόν εξέτασαν τα ζητήματα τα σχετικά με το με, το αίτημα του κυρίου Ζωάν Μαρί Ταγκαφόσο και του κυρίου Κρίστοφερ Στόκουελ. Τα δύο αυτά ε, ζητήματα ε, μας απασχόλησαν ε, καταρχήν από κοινού και μετά η Επιτροπή αποφάσισε να τα ξεχωρίσει. Όσον αφορά την αναφορά Ταγκαφόσο, οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί και εδώ υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών, εάν και κατά πόσον δηλαδή μπορούν να παρισφρήσουν στην ε, ε, δικαστική απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί όσον αφορά την δεύτερη αναφορά του κυρίου Κρίστοφελ Στόκουελ για την οποία είχαμε ζητήσει και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, αλλά και ζητήσαμε και γνωμοδότηση από την ε, Γιούρη, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ακούσουν του αναφέροντε ε, στην Ολομέλεια τη Επιτροπή και να αποφανθούν ε, περαιτέρω για την πορεία αυτή τη αναφορά, ε, λαμβάνοντα υπόψη και τις δύο γνωμοδοτήσει και τη νομική Υπηρεσία και τη επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αργότερα δεν θα δούμε κατά πόσο θα υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα κατά αυτήν την έννοια οι προτάσεις τώρα για αποστολές κατά το 2012 παρουσιάστηκε μία πρόταση ε, βάσει των ετοιμάτων που είχαν προωθήσει οι συντονιστές εξ ονόματος των μεμονωμένων ε, πολιτικών ομάδων και επί τη βάση του ειδικού βάρους που έχει ο κάθε συντονιστής επί τη βάση πάντα του καταλόγου που έχει υποβάλει η Γραμματεία ε, όσον αφορά το βάρος και το επί, τον επίγοντα χαρακτήρα των αναφορών και βεβαίως λαμβάνοντας ε, υπόψη και την αξιολόγηση των αποστολών που ήδη έχουν λάβει χώρα στο πρώτο τμήμα ε, της θητείας μας. Βάσει αυτών των στοιχείων και βάσει όλων των απόψεων των συντονιστών διετύπωσα ε, μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία ζητώ από το σύνολο της Επιτροπής ε, να δεχτεί ή να απορρίψει. Σας ζητώ λοιπόν να ψηφίσουμε επί της προτάσεως Μάλλον όχι. Πριν ψηφίσουμε έχουμε αιτήματα ομιλία. Η κυρία Όουκεν παρακαλώ. Δύο σχόλια. Βλέπω την ηλεκτρονική αλληλογραφία την οποία ανταλλάξαμε και είναι σαφές ότι και οι γκουε και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί είχαν ζητήσει την Ισπανία και την Ιταλία σαν τις δύο πρώτες ε, πρωτο, προτεραιότητές τους. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να... Ε, γιατί, γιατί θέλουμε να αναβάλουμε την Ισπανία. Ήταν σαφές βάσει της ηλεκτρονικής αλληλογραφία, την οποία εδώ έχω εκτυπώσει ότι θα πηγαίναμε σε αυτές τις δύο χώρες θα μπορούσα να προτείνω μια συμβιβαστική λύση, αν θέλετε να με ακούσετε βεβαίως. Ένα συμβιβασμό λοιπόν να προτείνω. Να αποφασίσουμε, να, συγγνώμη, να διατηρήσουμε αυτά που, και να εφαρμόσουμε αυτά που είχαμε αποφασίσει την προηγούμενη φορά, έτσι ώστε να κάνουμε τον Οκτώβρη στην Ισπανία αυτή την αποστολή, ενώ ταυτοχρόνως κάποιοι άλλοι θα πάνε στη Γερμανία. Οι δύο αποστολές δηλαδή να γίνουν ταυτόχρονα ε, και στην Γερμανία και στην Ιταλία με διαφορετική σύνθεση. Οι πληροφορίες που μας δώσατε καταδεικνύουν σαφώς ότι η Ισπανία ήταν πρώτη απόφαση και πρώτη επιλογή. Και αυτό φαίνεται καθαρά στα email και στις συζητήσεις μας. Δεν είχαμε αποφασίσει ε, άλλωστε να κάνουμε ψηφοφορία. Δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μια τέτοια ψηφοφορία και επομένω εγώ δεν πρόκειται να συμφωνήσω να υπάρξει τέτοια ψηφοφορία. Αν θέλετε να προχωρήσουμε με το συμβιβασμό που πρότεινα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να θέσω το εξή θέμα. Όχι, να μην αλλάξει αυτό για τη Γαλλικία, σύμφωνα με τη λογική μας εδώ της Επιτροπής Αναφοράν. Η επίσκεψη στη Γαλλικία τονίζεται σε τέσσερις αναφόρες ε, για την παρουσία εκεί από το 1999 ήδη μέχρι το 2010 ή 922 το 2010 για το Ρία Ντελβούργο στην Κορούνια 1322-2007 Ρία Φερόλ στην Κορούνια και πάλι η 260 1999 και 138 2009 του Ρίος Ντεβίγκο Τι γίνεται τα χρόνια αυτά ήρθαν ακριβώς αναφέροντες για να μας εξηγούν τι ακριβώς γίνεται εκεί με τους ποτάμια αυτά και με τις περιοχές αυτές όπου είναι οικοσυστήματα ιδιαίτερα σημαντικά και για την Ισπανία και για όλη την Ευρώπη και παρέμειναν ανοιχτές όλες οι αναφορές. Ήρθαν εδώ Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2010 και το Σεπτέμβριο του 2011 και πέρα από την απόφαση αυτή τους είχαμε πει ότι θα το μελετούσαμε να στείλουμε μια αποστολή ακριβώς εδώ σε όλες τις ομάδες όταν είπαμε ποιες ήταν οι προτιμήσεις μας, ποιες ήταν οι προτεραιότητες για τις επισκέψεις αυτές με εκπλήσει πραγματικά και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Χουντή τον συντονιστή που είναι απόν τώρα αλλά είπε ότι αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα η Γαλλικία και η κυρία από τους πράσινους είπε και ευκίνη ότι ήταν πρώτη προτεραιότητα η Γαλλικία και σοσιαλιστές δεύτερη προτεραιότητα ε, και ο Σαλαβράκο η ομάδα του ε, πρώτη προτεραιότητα και από τους ελεύθερους ε, πρώτη προτεραιότητα. Άρα λοιπόν πέρα τώρα από τη λογική της ομάδας υπάρχει μια άλλη λογική που θα πρέπει να υπερισχύει των άλλων. Είναι η λογική των αναφερόντων. Έτσι. Και οι υπόλοιπε ακολουθούν τώρα. Εάν ψηφίσουμε τελικά, τι θα ζητούσα να είναι σαφές ε, ότι η Επιτρο... το ταξίδι αυτό έτσι και ε, τουλάχιστον εγγυημένα θα γίνει το 2013 για να δώσουμε μια απάντηση σε αυτές τις περιοχές ε, στη Γαλλικία και ακριβώς στα φιόρντ και στις εκεί περιοχές και να μπορέσουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε υπέρ Βέβαια του να ήταν αυτή τη χρονιά, αλλά προσφέρουμε την εγγύηση ότι τουλάχιστον το 2013 θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι αυτό, η επίσκεψη αυτή εκεί. Η Μιράντα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι ο κύριος στόχος αυτών των αφορών ήταν ακριβώς η βάση τους. Ήταν ε, να εξηγιάνουμε αυτά τα ύδατα. Έτσι, έτσι πέρα τώρα από την κυβέρνηση υπάρχει μια ε, διαδικασια επιπαραληψη παραλήψη. Υπάρχει ένα κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν μπορούν να εργαστούν εκεί. Γιατί ακριβώς τα ύδατα εκεί, στα φιόρντα αυτά της Γαλλικίας και στο Βίγκο και στο Φερόλ και στην Κορούνια δεν ε, έχουν καθαρίσει γιατί δεν ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις μας ακριβώς. Όταν εδώ ε, βλέπουμε εδώ και στη Γερουσία ότι ανέλαβαν την υποχρέωση όταν κυβερνούσαν να, το, να τα καθαρίσουν αυτό ακριβώς και ότι θα το έκαναν και η προηγούμενη κυβέρνηση και θα χρωστάμε μια απάντηση, μια εξήγηση. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Άρα λοιπόν το να αναβληθεί σημαίνει ότι τους κοροϊδεύουμε, τους δουλεύουμε το να την πάμε σαν προμηνία σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε αυτά που υποσχεθήκαμε σαν ομάδες ε, και ανάμεσα αυτούς και στους σοσιαλιστές και ζήτησαν τη βοήθειά μας οι πολίτες οι αναφερόμενοι. Θα πρέπει εκεί να μεταβεί μια αντιπροσωπεία. Ε, θα, θα ήταν αρνητικό να μην πραγματοποιηθεί τελικά αυτή η επίσκεψη. Ο Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Μιράντα, αυτό ακριβώ ότι κοροϊδεύει κανείς κάποιον είναι ότι να σκέφτεται, να, να επισκέπτεται μια φορά την άλλη. Αυτά, σε αυτή τη θητεία πόσες ε, ε, αναφορές ήρθαν από 27 χώρες και πώς επισκεφθήκαμε 6 χώρες και μια από αυτές ήταν και η Ισπανία και θέλετε να επιστρέψουμε στην Ισπανία 21 άλλες χώρες εκεί καμία εμφάνιση δεν πήγαμε που δεν είναι γιατί πάντα έτσι στην Ισπανία γιατί στην Ισπανία επαναλαμβάνω εδώ πέρα από το περιεχόμενο κυρία Μιράντα αυτό ακριβώς για την Επιτροπή Αναφορών. Δεν μπορεί να είναι η Επιτροπή Αναφορών που θα ασχολείται μόνο με τα ε, ισπανικά θέματα και την κυρία Θα πρέπει να είναι μια Επιτροπή Αναφορών που να μην ασχολείται με μια και μόνο χώρα. Γι' αυτό ακριβώς ε, αυτή η τοποθέτηση, όπως σας το είπα και εγώ στο περιεχόμενο εδώ, δεν έχει σχέση με αυτό. Εδώ εντάξει θα μπορούσαμε να τους εγγυηθούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι που έχουν, παραμένουν ανοιχτές οι αναφορές τους και περιμένουν επίσκεψη. Έχουμε ουρά ολόκληρη που κάνουν και πολλές άλλες αναφορές πολύ πριν από τους συμπατριώτες σας από τη Γαλλικία. Έτσι κυρία Πρόεδρε. Ναι, εσείς καν υποβάλατε μια πρόταση και εγώ υπέβαλα το πεσήμα το πρωί όπως είχε ο κ. Μέγερ. Εντάξει εδώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα δούμε την επόμενη χρονιά, θα δούμε και υπόλοιπε χώρε. Γιατί, επιμένω, για ρίξτε μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα. Πόσε φορέ πήγαμε στη μια χώρα και πόσε φορέ πήγαμε σε άλλε χώρε. Ακούστε, εδώ δεν είναι να σεβαστούμε ένα χρονοδιάγραμμα, όχι. Εμεί δώσαμε ένα λόγο. Το Οκτώβριο το κάναμε αυτό. Έτσι. Και εδώ δεν είναι τίποτα κατά ενό κράτου μέλου. Είναι για να σεβαστούμε αυτά που είπαμε. Μιλάει ταυτόχρονα ο κ. Στρογγάη. Ναι, η κυρία Μιράντα δεν ζήτησε καθόλου το λόγο και όμως ε, μιλάει από μόνη της, λέει ο κ. Σατρογκάης. Όντως, υπάρχει και δυσκολία άλλωστε όταν μιλά το ένας πάνω στον άλλον, ούτε οι διερμηνείς δεν μπορούν ε, να μεταφράσουν και είναι ανώφελη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, λυπούμε αγαπητοί συνάδελφοι γιατί ξαναρχίζουμε τέτοιου είδους ε, συζητήσεις. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αφορά απλά διαδικαστικά θέματα οργάνωσης των εργασιών. Το γεγονός ε, της ε, αναπομπής ε, ή αλλαγής κάποιας σειράς των αποστολών δεν σημαίνει ότι αποδίδεται μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία στη μία ή στην άλλη χώρα, στη μία ή στην άλλη αποστολή. Επίσης, δεν πρέπει να καταλογίζονται προθέσεις από τις ενδείξεις που έλαβα από τους ε, συντονιστές, εγώ εκπώνησα μία πρόταση, έκανα μία ε, πρόταση για συγκεκριμένες αποστολές ε, και βασίστηκα σε ενδείξεις και σε πληροφορίες που μου έστειλαν όλοι οι συντονιστές, χωρίς κάποια σειρά προτεραιότητας. Όμως εγώ οφείλω να σημειώσω, να λάβω υπόψη μου το πολιτικό βάρος του κάθε συντονιστή. Είπαμε ότι μπορεί να γίνει η αποστολή, η επίσκεψη στην Ισπανία ε, στις αρχές του 2013 και τώρα να αποφασίσουμε για το 2012. και όπως έχει ζητηθεί και από κάποιους ε, συντονιστές, γιατί έχω λάβει διάφορα ε, mail τα οποία μπορώ να σας ε, στείλω να τα διαβάσετε αν θέλετε. Η αποστολή στη Γαλλικία μπορεί ωραιότατα να λάβει χώρα στην αρχή του επόμενου έτους, το 2013 και δεν νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στα συμφέροντα των πολιτών. Ε, άλλωστε υπάρχει και μια διαδικασία επιπαραβάση η οποία δεν ολοκληρώνεται, ε, άρα ωραιότατα μπορούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε από κοντά όλες τις διαδικασίες, όλες τις κατηγορίες οι οποίες αφορούν την περιοχή αυτή και να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτού του θέματος. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε την πρόταση έτσι όπως έχει διατυπωθεί, διότι πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνεται ορθώς ε, και αυτή η συμβαστική πρόταση του συναδέλφου Μάγερ. Ε, δηλαδή να αναφέρω ρητά ότι αυτή η αποστολή στη Γαλλικία μπορεί να γίνει στην αρχή του 2013 και θα είναι η πρώτη αποστολή του επόμενου έτους. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε επί αυτής ε, της προτάσεως έτσι όπως έχει υποβληθεί υπέρ της προτάσεως κατά, κατά, αποχές, Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 13 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και 4 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η πρόταση έτσι όπως αρχικώς υπευλήθη. Οι οι συντονιστές επίσης ενέκριναν την πρόταση ημερήσιας διάταξης με τις τροποποιήσεις σχετικά με, τις, με την αναφορά ταγκαφός όπως είπα προηγουμένως και επίσης ενέκριναν την απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί μετά το πέρας της εξέτασης των ε, αναφορών για την κακή μεταχείριση των ζώων και απεφάσισε λοιπόν ε, να ε, υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτοιμα για προετοιμασία πρότασης ψηφίσματος. Θα ζητούμε λοιπόν, θα υποβάλουμε αυτό το αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν λήφθησαν άλλε αποφάσει στη διάρκεια τη συνεδρία των συντονιστών και επομένω κλείνουμε το σημείο αυτό της μερισίας διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ε, εξέταση των αναφορών που έχουν εγγραφεί εις το πρόγραμμα της απογευματινής συνεδρίασής μας. Έχουμε παριστάμενους ε, αναφέροντες οι οποίοι θα πάρουν το λόγο στη διάρκεια των εργασιών. η Πρώτη αναφορά εγγεγραμμένη στη μερίσια διάταξη είναι η παριθμόν 886 του 2011 που έχει υποβάλει ο Βέσκο Ντίμοβ και που συνοδεύεται από περίπου 8.000 υπογραφές πολιτών και που θα εξεταστεί μαζί με την 1378 ε, του Θείοντορ Ουρμπανόβιτς.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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Βάσκο Ντίμοβ και έρχομαι από τον Άβη Μπαζένα. Δέκα μήνες πριν οργανώσαμε στον Νόβι Μπαζάρ μια ε, επιτροπή στόχος της οποίας ήταν ε, να ε, ενενδιωθούμε στην απόφαση της βουλγαρικής κυβέρνησης να δώσει άδεια στην Αμερικανικών των Σευρών εταιρεία έτσι ώστε να προχωρήσει σε εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Το Νόβι Μπαζάρ είναι μια μεγάλη περιοχή και ε, οι έρευνες θα έλαβαν χώρα ακριβώς αυτήν. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή ε, υπάρχουν σημαντικά ιστορικά ε, μνημεία ε, και ε, πρόκειται στη, για ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ε, μνημείο το οποίο είναι μοναδικό στη Βαλκανική Χερσόνησο. Πρόκειται για μια, ε, για μια περιοχή η οποία είναι ε, πολύ επίπεδη, ιδιαίτερα έφορη, χωρίς ε, πηγές, χωρίς ιδιαίτερα σημεία νερού. Το, η μόνη πηγή βρίσκεται σε πολύ χαμηλά στρώματα ο υδροφόρος ορίζοντας δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Επομένως, ε, η πραγματοποίηση ερευνών ε, είχε ξεκινήσει ε, παλαιότερα για προσπάθεια εξέβρεσης πετρελαίου. Εδώ βλέπετε μία δεξαμενή ε, νερού ε, σαν αυτές που βλέπει κανείς συχνά στην περιοχή αυτή. Στο πάνω μέρος βρίσκεται η δεξαμενή από την οποία παίρνουν νερό ε, οι περισσότερες πόλεις της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας έχουν χτιστεί οι δεξαμενές αυτές γιατί όπως είπα δεν υπάρχει η φυσική ροή το, του εδάφους σε λήψη πρανών. Έχουμε συλλέξει 8.000 ε, υπογραφές ε, και είδαμε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαμε πολύ μεγάλη στήριξη. Είναι σαφές ότι η περιοχή αυτή υποφέρει από λειψιδρία και επομένως πρέπει, είναι σαφές ότι πρέπει να κατεβούμε στα 150 έστω και 200 ακόμα μέτρα ε, στον υδροφόρο ορίζοντα για να βρούμε νερό. Γι' αυτό λοιπόν ε, ξεκίνησε ένα κύμα διαμαρτυριών σε πολλές πόλεις ε, της περιοχής με συμμετοχή πολλών νέων, νέα, οικογενειών με μικρά παιδιά γιατί όλοι φοβούνται ότι θα δηλητηριαστεί, θα μολυνθεί το νερό της περιοχής. Ε, η περιφέρεια, η περιοχή μάλλον όπου θα γίνουν αυτές οι ερευνές ε, καλύπτουν περίπου το 1 τέταρτο του ε, εδάφους της Βουλγαρίας όπου ζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές. Αυτά είναι, αυτός είναι ο προβληματισμός μας. Θέλουμε καθαρό νερό, θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το γόνιμο έδαφος της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Madam Chairman, just a few sentences. As I would like to welcome you. Πρόεδρος. Θα ήθελα την πρώην συνάδελφο να χαιρετήσω, η οποία και προωθεί την πρωτοβουλία αυτή και που η ίδια έζησε σαν μέλος του Κοινοβουλίου και σαν μέλος της Επιτροπής μας τα πράγματα. Η κυρία Βράτκοβα, με συγχωρείτε το πως προφέρω το όνομά σας, σας δίνω το λόγο πάντως, με κάθε καλή διάθεση. Πολύ λίγα, κυρία Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λίγα θέλω να προσθέσω. Παρά το ότι η Βουλγαρική Βουλή ψήφισε ένα μορατόριο για την ε, έρευνα και εξόριξη σχιστολιστικού αερίου υπάρχει ο κίνδυνος γιατί μια νέα επιτροπή ad hoc συστάθηκε πρόσφατα και κατά πάσα πιθανότητα θα αποφασίσει να επανεξετάσει το ζήτημα και να αναθεωρήσει την απόφαση. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία και θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των Ευρωβουλευτών και να κάνουμε έκκληση να παλέψετε μαζί μας. Όχι μόνο η φύση στη Βουλγαρία, αλλά και η φύση και το μέλλον των παιδιών μας. Η φύση και το μέλλον της Ευρώπης εξαρτώνται. Πρέπει όλοι μαζί να πούμε όχι στην έρευνα και εξόριξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Κάτι ακόμη. Έχω εδώ ένα χάρτη. Στο χάρτη εδώ είναι σαφές ότι η Βουλγαρία δεν έχει μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου από αυτή την πηγή. Δεν έχει καμία έννοια να ξεκινήσει η εκμετάλλευσή του. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Το ρόλο έχει τώρα ο Φλωρέντης Λιμέα από την Επιτροπή. Η Φλωρέντς. Ευχαριστώ. Μετά την ε, υποβολή της αναφοράς, η Επιτροπή έστειλε ένα επίσημο αίτημα στις βουλγαρικές αρχές για πληροφόρηση όσον αφορά τη συμμόρφωση του προγράμματος με τον ε, ενωσιακό περιβαλλοντικό νόμο και ιδιαίτερα με την οδηγία για την έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόσφατα λάβαμε τη βουλγαρική απάντηση, την οποία εξετάζει η Επιτροπή, οι υπηρεσίες μας, και θα τη συζητήσουμε περαιτέρω με τι βουλγαρικές αρχές. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα τηρήσει ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα περαιτέρω βήματα που θα ληφθούν. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση. Η συνάδελφος Κολάσκα Μπομπίνσκα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για το δημιουργικό φυσικό αέριο ε, και για τον, ε, ε, για τον κίνδυνο ανάλυσης των δεδομένων. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι κίνδυνος αυτό. Είναι πολύ καλό να προστρέχει κανείς τα στοιχεία, είτε πρόκειται για μια επιτροπή, είτε για ένα όργανο και να ξανααναλύει τα στοιχεία. Η κίνηση στη Βουλγαρία ήταν ε, αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών αποφάσεων, κάποιων διαμαρτυριών, ε, διότι η απόφαση δεν είχε βασιστεί σε πραγματικά στοιχεία ε, και σε δεδομένα. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή εξέλιξη πρέπει να σκεφτούμε όχι μονάχα τι μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά και ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνονται. Ε, για την Πολωνία ας πούμε το σχιστολιθικό φυσικό αέριο είναι πολύ καλό γιατί μας δίνει την δυνατότητα ενεργειακής αυτάρκειας. Ε, το σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα καλού ενεργειακού μείγματος ε, σε κάθε χώρα. Εάν η Επιτροπή αποφανθεί ότι δεν ε, παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, ότι ε, ακολουθούνται ορθά ε, οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος, τότε αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί θα είναι το σωστό ενεργειακό μείγμα. Και άλλωστε αυτό είναι και το αίτημα της επόμενης της πολωνικής αναφοράς που ακολουθεί. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για να τα πω τώρα. Είναι ευρωπαϊκής φύσης το πρόβλημα. Από το συμπέρασμα θα ξεκινήσω. Ναι, από τη στιγμή οι πολίτες, οι Βούλγαροι μας απευθύνονται σε εμά, αλλά και οι Πολωνοί. Και θα έχουμε νέα αναφορά στην Επιτροπή Αναφορά από τους Γάλλους πολίτες για το σχιστολιθικό αυτό φυσικό αέριο. Έχουμε τουλάχιστον τρία κράτη, τους πολίτες από τρία κράτη τα οποία απευθύνονται σε εμά. Άρα λοιπόν αποκτά το θέμα μια κάποια νομιμότητα εδώ ακριβώς γιατί για την εκμετάλλευση αυτού του αερίου βλέπουμε στα πλαίσια αυτά σήμερα αποτελεί ευρωπαϊκό θέμα και από τη στιγμή που απευθύνονται σε εμά, νομίζω ότι επισέρχονται στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Θα ολοκληρώσω και θα ήθελα έτσι άμεσα και να απαντήσω. Ε, τι μας ζητείτε στα πλαίσια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Το θέμα μιας εκτίμησης εκτίμησης επιπτώσεων από την εκμετάλλευση, ή την εξόριξη αυτού του αερίου στη Βουλγαρία κυρίως και μάλιστα σε, ε, με ειδικά τοποδικές συνθήκες όπως μας είπε αναφέρον δηλαδή ιδιαίτερα γόνιμη περιοχή έτσι στο υπεδαφός της ήδη και που είναι ιδιαίτερα εύθραυστη περιοχή όσον αφορά την εξέβρεση ύδατος και ακριβώς ε, μετά από όσα είδαμε στις Ηνωμένε Πολιτείες και με διάφορες μελέτες, η εξόριξη εκμετάλλευση αερίου προκαλεί πολλά προβλήματα ακριβώς πώς θα διαφυλαχθούν οι πηγές ύδατος. Έτσι. Και αυτό που ζητείτε είναι μια εκτίμηση, μια μελέτη επιπτώσεων και ο συνάδελφος εδώ θα λάβει το λόγο γιατί στην Επίτροπη Περιβάλλοντος θα έχουμε μια έκθεση σχετικά με το αέριο και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε αυτή την ανέλυση ότι χρειάζομαστε ακόμα κάποιες εκτιμήσεις επιστημονικής φύσεως και θα πρέπει να δούμε σε κάθε περίπτωση ακριβώς μια μελέτη ε, επιπτώσεων πριν οποιαδήποτε εξόριξη εκμετάλλευση και ακόμα κάτι για τις επιπτώσεις επειδή βήμα-βήμα προχωράμε γιατί απαιτείται μια προκαταρτική μελέτη και η εφημερίδα Libre μας λέει για μια νέα μελέτη από την ε, αρμόδια περιοσία, υπηρεσία της ε, των ΗΠΑ για την εκμετάλλευση ακριβώς και ότι υπάρχουν μικροσυσμοί ακριβώς επειδή υπάρχουν, ε, υπάρχει μια αστάθεια στο υπέδαφος μετά λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και σας λέω ότι σκέφτομαι ότι ε, το ότι απευθύνθηκαν σε εμά είναι κάτι το κανονικό, έτσι. Και θα πρέπει και η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε και των Πολωνών πολιτών παρόμοια αναφορά και των Γάλλων σε λίγο. Θα ήθελα να προτείνω να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, να οργανώσουμε μια ακρόαση με όλους αυτούς που επιβάλλουν αυτές τις αναφορές, ίσως προσθεθούν και άλλοι και στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής να οργανώσουμε την όλη συζήτηση για το τι γίνεται σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο και πώς θα ανταποκριθούμε, πώς θα απαντήσουμε στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών, εκείνων που απευθύνονται σε εμά την Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Sonic. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ο μιλήτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αύριο στις 11 το πρωί θα παρουσιάσω ε, την έκθεσή μου σχετικά με το σχιστολιστικό φυσικό αέριο και την επίπτωσή του στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό ε, δείχνουμε και στους αναφέροντες ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά, που μας ενδιαφέρει ε, και ε, το συζητάμε άλλωστε ε, και ο Επίτροπος Χέντιγκερ ανέφερε ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή πηγή ενέργειας για την Ευρώπη και, και βεβαίως θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι πρόνοιες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος αυτό είναι σαφές και να ληφθούν υπόψη όλες οι μελέτες. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ε, μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι ε, οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι ικανές να προστατέψουν το περιβάλλον. Ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε περιπτώσεις προβλήματος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για την περίπτωση του αμίαντου ας πούμε, φέρθηκε με σωστό τρόπο. Εδώ βέβαια αναφερόμαστε στην εξόριξη και την εκμετάλλευση ε, ε, μιας πηγής ενέργειας ε, και για την ώρα δεν έχουμε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Ξέρουμε βεβαίως ότι στην ε, Ευρώπη λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται. Θέλουμε, ε, η κάθε χώρα βεβαίως θέλει να προστατέψει το περιβάλλον της ε, και θα πρέπει και η κάθε χώρα μόνη της να αποφασίσει μέχρι που θέλει να φτάσει όσον αφορά την εκμετάλλευση του και την εξόριξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Ε, ξέρουμε ότι στην Βουλγαρία ε, η διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό μάλλον δεν έγινε πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστεί πρώτα απ' όλα η κοινή γνώμη ότι όλα γίνονται με τρόπο ορθό και διαφανή. και βεβαίως αυτό δεν αφορά μονάχα το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, αφορά και όλες τις άλλες επιλογές ενέργειας ε, και ε, επίσης εσείς αναφερθήκατε σε 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε και για μεγαλύτερες περιοχές και για μεγαλύτερες γεωτρήσεις, ενώ γεωτρήσεις που φτάνουν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, μέχρι και τα 500 ε, μέτρα θα πρέπει να μελετήσουμε όλες αυτές τις μορφές εξόριξης έτσι ώστε να γνωρίζουμε σαφώς ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι είναι ε, ασφαλής οποιαδήποτε μορφή εξόριξης. Ευχαριστώ η κυρία Γιώτοβα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μπέγε και στηρίζω την πρότασή της να γίνει μια ακρόα στην Επιτροπή μας για τα θέματα του αερίου αυτού και όλων αυτών των αναφορών. Και θα συνεχίσω στα βουλγαρικά σεβόμενοι τους ε, βούλγαρους παρόντες. Είμαι κατά της ε, έρευνας και εξόριξης σχιστολιθικού αερίου. Στις 16 Ιουνίου 2011 η κυβέρνηση υπέγραψε μια σύμβαση με την Αμερικανική εταιρεία Chevron για να ερευνήσει και να εξορίξει σχιστολιθικό αέριο στο Νόβι Παζάρ, στο μπλοκ 1. Αυτό συμπεριλαμβάνει διάφορες μεγάλες ε, πόλεις, είναι ο Σιτοβολώνας της Βουλγαρίας και πολλές, ε, πολλά αποθέματα ε, ποσίμου ύδατος. Μετά τις αναλύσεις που έκαναν οι περιβαλλοντολόγοι σε μια περιοχή που είναι το 1 τρίτο της Βουλγαρίας και πάνω από 90% της βορειοανατολικής Βουλγαρίας θα είναι αντικείμενο έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Επειδή όμως ε, η γη, τα εδάφης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και επειδή για αυτήν την ε, υδραυλική διερεύνηση χρησιμοποιούνται κάποια χημικά που δεν ξέρουμε καν ακριβώς ποια είναι γιατί η εταιρεία που τα χρησιμοποιούν ε, θεωρούν και μας λένε ότι είναι εμπορικά μυστικά. Ορισμένα όμως είναι ιδιαίτερα τοξικά. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξοριχθεί αυτό το αέριο. Υπάρχει λοιπόν πολύ ισχυρή διαμαρτυρία κατά της ε, έρευνας για το αέριο αυτό. 70.000 έχουν υπογράψει κατά αυτής της εκμετάλλευσης και αποκαλούν το κίνημά τους εναντίωση σε ένα βουλγαρικό Τσερνόμπιλ. Έχουν γίνει χιλιάδες ε, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στη Βουλγαρία κατά αυτής της προσπάθειας και δεν συμφωνώ με την κυρία Μπομπίνσκα από την Πολωνία διότι πρώτον πρέπει να σεβαστούμε τη γνώμη των πολιτών ανεξάρτητα από το εμπορικό κέρδος που μπορεί να προκύψει. Μετά τις ε, διαμαρτυρίες ε, στη Βουλγαρική Βουλή ψηφίστηκε ένα μορατόριο, αλλά είναι κάτι το προσωρινό. Στόχος του μορατόριου ήταν αρχικά να υπάρξει περισσότερη συλλογή στοιχείων για το πώς θα γίνει η έρευνα και η εξόριξη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Υποπτευόμαστε μάλιστα ότι δεν έχουν ε, γίνει αυτές οι μελέτες γιατί θα μπορούσαν να καταδείξουν ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Ότι δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα του περιβάλλοντος της χώρας μας θα καταστραφεί. Οι συνάδελφοι από τη Ρουμανία ξέρω ότι υπήρξε εκεί μια συμφωνία για το σχιστολιθικό ε, αέριο αλλά αυτές οι μελέτες και η εξόριξη θα γίνουν πολύ κοντά στα βουλγαρο-ρουμανικά σύνορα, μόλις ένα χιλιόμετρο. Κατηγορηματικά δηλώνω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, και να τους καταγγείλω μάλιστα, διότι ε, ήρθαν εντελώς απροετοίμαστε εδώ πέρα. Μας είπαν ότι ακόμη περιμένουν για περαιτέρω απαντήσεις από τις βουλγαρικές αρχές. τι είδου άποψη είναι αυτή της Επιτροπής. Με βάση ανεπίσημες πληροφορίες που έχω πάρει ως ε, Ευρωβουλευτής από τη Βουλγαρία, μόλις πριν από μια ώρα η βουλγαρική κυβέρνηση πρόκειται να διακόψει αυτό το μορατόριο παρά το ότι το ψήφισε η Βουλή. Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος για να τηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Okay. Θα είμαι σύντομη. Φυσικά υποστηρίζω περαιτέρω προσπάθειες για να γίνει μία ακρόαση, να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Καλό την Επιτροπή. Εάν το θέμα είναι εάν έχει γίνει οποιαδήποτε έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης φέτος. Έχουμε και την ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Και ίσως να καλύπτεται και το πρόγραμμα REACH. Δεν είναι καινοτόμο τρόπος αυτός που σκέφτεστε. Δεν λαμβάνει υπόψη τα θέματα της αλλαγής κλίματος. Βεβαίω, είναι η πολιτική μου αποτίμηση αυτή. Κοιτάξτε, έχω πέντε γόνια. Για, για μένα ε, είναι ζωτικό να κάνουμε κάτι για το μέλλον τους και για τα παιδιά των εγγονιών μας, τα δυσέγγονά μας. Αυτά που κάνουμε, αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών, καθώς και όσα συμβαίνουν για την ε, οδηγία, για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, όπου ε, ναι μεν εγκρίναμε ένα πολύ καλό ψήφισμα, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά κράτη-μέλη που σκέφτονται μαύρα θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή ακριβώς η συνάδελφος Γιώτοβα μόλις είπε ότι η κυβέρνηση κατέληξε συμφωνία με τη Σεύρον. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν να μου πει η Επιτροπή πόσο έχει επενδύσει φέτος η Σεύρον. Γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν κατηγορώ ότι δώρο δόξαν κανένα. Αλλά ε, όταν ε, υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει κανείς πολλά λεφτά, το έχω δει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, τα χρήματα μπορεί να είναι πολύ πιστικά και πολύ αποτελεσματικά. Ακόμη και είναι αποτελεσματικά σε μια βλακώδη προσπάθεια να καταστρέψουμε το περιβάλλον. Σας παρακαλώ να μου πείτε πόσα χρήματα έχουν ήδη δοθεί για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις αναφορές αυτές, τονίζοντας ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην έρευνα και την εμπορική εκμετάλλευση. Ας μάθουμε από τα λάθη των άλλων. Αυτό που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνονται μεγάλες κλίμακας εμπορικές ανασκαφές και βλέπουμε τι ζημιά δημιουργείται στα ύδατα. Βλέπουμε τι ζημιά δημιουργείται λόγω της πρόκλησης μικροσυσμών. Βλέπουμε τη ζημιά που υπάρχει στην υγεία των ανθρώπων. Βλέπουμε ασθένειες ε, στα ζώα υποτίμηση της τιμής των ακινήτων και, των, ε, και της γης. Απειλούνται ζωές και εισοδήματα. Πριν λοιπόν ε, και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσουμε παρόμοια τακτική, ας μάθουμε από τα παραδείγματα αυτά. Ας μην ξανακάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι. Ας μην ορμήσουμε με το κεφάλι μπροστά γιατί θεωρούμε ότι είναι επικερδής δραστηριότητα. Νομίζω ότι είναι θέμα ενωσιακής αρμοδιότητας. Το μισό μας χρόνο μιλάμε για την ανάγκη μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Και στην πραγματικότητα εξάγουμε φυσικό αέριο από το μεθάνιο, έχουμε την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος λέγοντας ότι πρέπει ο άνθρακας που προκαλείται από αυτή την εξόριξη να συλλαμβάνεται. Και έχουμε την εταιρεία Tindel στο Ηνωμένο Βασίλειο που τονίζει την πολύ σοβαρή εταιρεία αυτή ε, συμβουλών για το περιβάλλον που μας λέει ότι ο καλύτερος τρόπος για να ε, αξιοποιηθεί το σχιστολιθικό αέριο είναι να παραμείνει κάτω από το έδαφος. Διότι αν το βγάλουμε στην επιφάνεια θα έχουμε τρομερές εκπομπές άνθρακα πολύ σοβαρότερες αρνητικές επιπτώσεις από την αποδοτικότητα αυτού του ενεργειακού πόρου. Ας μάθουμε λοιπόν από την πείρα των άλλων, ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την αλληλοκατανόηση των ενωσιακών θεσμών, ας κάνουμε μια ακρόαση ούτω ώστε να αισθανθούν και οι αναφέροντες ότι λαμβάνονται υπόψη και υποθέτω ότι θα έχουμε και αναφορές και από τον Ομένο Βασίλειο για το θέμα αυτό. αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να κανονίσουμε ακροάσεις και να μοιραστούμε πληροφόρηση. Θα ήταν ανόητο επειδή η Σεύρον δίνει δισεκατομμύρια να τις δώσουμε τη δυνατότητα εξόριξης ή να είμαστε πιο έξυπνοι, να σκεφτούμε τα πέντε γκόνια τη κυρία Όκεν, τα τρία δικά μου, να σκεφτούμε τα δικά τους συμφέροντα και το μέλλον τους, να είμαστε επιφυλακτικοί. Και βασίζομαι σε εσά Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να δηλώσω εξ αρχής ότι είμαι κι εγώ ο παππούς. Ε, και με ενδιαφέρει, και έχω και ανήψια και με ενδιαφέρει ποια Ευρώπη θα, παραλάβουν, θα παραδώσουμε μάλλον εμείς ε, στην επόμενη γενιά. Έχουμε εδώ μία αναφορά από τους Βούλγαρους ε, φίλους, συναδέλφους ε, και γείτονες, αλλά είναι déjà vu. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες έγινε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση όσον αφορά τις προθέσεις της ρουμανικής κυβέρνησης να δώσει συμβόλαιο στην ίδια Αμερικάνικη εταιρεία για την εξόριξη και την ε, εκμετάλλευση στην Ανατολική Μολδαβία, κοντά στον Περλάτ και επίση άλλη μία στην Τομπρόζα, κοντά στην, ε, στα βουλγαρικά σύνορα. Δύο αδειοδοτήσεις λοιπόν. Για να καταλάβετε δε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας και πόσο σημαντικό είναι να γίνει ευρωπαϊκό ζήτημα, να σας πω το εξή. Γιατί εγώ μιλάω για πράγματα που τα ξέρω. Στην ε, περίπτωση της Ρουμανίας η κυβέρνηση ουδέποτε υπέβαλε ΕΠΕ ενώ έδωσε την αδειοδότηση για την εξόριξη και την εκμετάλλευση του αερίου. Κανείς, ούτε ο Πρωθυπουργό, ούτε οποιοδήποτε υπουργό, ούτε καν ο Υπουργό Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην τεράστια ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης και καλής αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Υπάρχουν ε, ε, ζητήματα τα οποία αφορούν τη γεωργία, ε, τις μικροτεκτονικές τεκτονικές κινήσεις, την μόλυνση των υδάτων κτλ. Αναφέρεται σαφώς ο αυξημένος κίνδυνος ρογματώσεων του εδάφους και μικρών σεισμών δεν υπήρξε καμία διαφάνεια, όπως άλλωστε και στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Ουδέποτε, είτε η κυβέρνηση, είτε οποιαδήποτε δημόσια αρχή προχώρησε σε οποιοδήποτε δημόσιο διάλογο με τις αφορόμενες περιοχές. Ποτέ δεν έγινε συζήτηση σε οποιοδήποτε κοινοτικό γραφείο του, του Μπερλάτ με τόσους κατοίκους. Ποτέ σε έστω Δημαρχείο δεν έγινε μία συζήτηση, έστω και αν υπήρξαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Πολλό δε μάλλον η ρουμανική κυβέρνηση, χωρίς να υποβάλει οποιαδήποτε πληροφορία για τη σύμβαση, ε, το κατέγραψε ως ε, απόρριτο στοιχείο. Καταλαβαίνετε για ποια διαφάνεια μιλάμε. Τέλος, εάν εμείς οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι ας πούμε ότι είμαστε ανόητοι. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Τότε γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε πρόσφατα να αναβάλει οποιαδήποτε εξόριξη της, του αερίου αυτού. Γιατί και η Γαλλία αποφάσισε αποφάσισε να απορρίψει για την ώρα και να απαγορεύσει την ε, εξέλιξη, ε, ε, συγγνώμη, την προώθηση των ερευνών. Γιατί δύο ηγετικές χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη και την έρευνα αποφασίζουν να σταματήσουν ε, και επομένως ε, γιατί άλλες να αποφασίζουν να ε, ενστερνιστούν τόσο επικίνδυνες τεχνολογίες θέτοντας σε κίνδυνο όλους τους ανθρώπους, τις κοινωνίες που ζουν εκεί, χωρίς και μια σωστή επιχειρηματολογία που θα αποτελεί βάση αυτής της απόφασης. Προτείνω λοιπόν να έχουμε την ακρόαση, να αφήσουμε ανοιχτές τις αναφορές Θυμηθείτε αυτό που σας είπα, ότι κι άλλες χώρες θα προσθεθούν σε αυτή τη λέσχη των τεσσάρων χωρών που έχουν ήδη υποβάλει αναφορές. Θα υπάρξουν οπωσδήποτε και Ρουμάνοι ε, οι οποίοι θα προχωρήσουν με υποβολή κάποιας αναφοράς γιατί είναι πολύ ε, αντίθετοι με τη διαδικασία αυτή και επομένως ε, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει αυτή τη φορά πια να βρεθούμε και μπροστά σε τελεσμένα γεγονότα. Θα πρέπει να ε, αντιδράσουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε νεκροψία στην περιοχή, θέλουμε να προστατέψουμε την περιοχή. Είναι ουσιώδους ε, σημασίας οι κύριες οδηγίες να εφαρμοστούν, να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη ε, να ε, εφαρμόσουν σωστά τους υφιστάμενους ε, κανονισμούς και την υφιστάμενη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Κανείς άλλος δεν έχει δει τον λόγο. Μήπως η Επιτροπή θα μπορούσε να απαντήσει. Στο τέλος, το τέλος. Εσείς. Η Επιτροπή μήπως θα μπορούσε να προβεί σε μια κάποια διευκρίνηση. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ή εκπρόσωπος. Να διευκρινίσω τι ακριβώς κάνουμε γιατί δεν φαίνεται να το γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής σας. Πρώτα απ' όλα έχουμε δώσει βοήθεια όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωνικού κεκτημένου. Υπάρχει η οδηγία για τις ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ένας γιατρός, ήταν ένα γιατρό πίσω. Sorry, Μισό λεπτό, περιμένουμε για πέντε λεπτά και ένα γιατρό, έτσι. Ε, ελπίζω να συναντήσω την κατανόησή σας.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Κοίτα και να γίνεις Δυστυχώς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 Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Good luck for the young lady who fainted. Ε, λιποθύμησε μία κοπέλα. Συγγνώμη, αλλά ήταν αναγκαίο να διακόψουμε. Νομίζω ότι είχε η εκπρόσωπος της Επιτροπής το λόγο. Ήθελα να διευκρινίσω τις δραστηριότητες μας για να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν από πλευράς ε, κάποιων ευρωβουλευτών. Όπως ήδη υπόθηκε, η Επιτροπή έχει δώσει οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτή, η, αυτό το κείμενο είναι προσβάσιμο στο ίντερνετ. Επίσης η Επιτροπή έχει παραγγείλει μια σειρά από μελέτες για να συλλέξει πληροφορίες για τους ενδεχόμενους ε, περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις από αυτήν την ε, διαδικασία υδραυλικής ρογμάτωσης σε συνδυασμό με οριζόντια εξόριξη. Περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε τα αποτελέσματα. Και όσον αφορά τις εκκλήσεις αερίων θερμοκηπίου, έχουμε ζητήσει μέσω της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική Δράση μια άλλη λοιπόν έρευνα που περιμένουμε να μας υποβληθεί τον Ιούνιο τρέχοντος. Επίσης ε, κοιτάμε και τις σωρευτικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν ιδιαίτερα για τον υδροφόρο ορίζοντα και τη χρήση της γης στην Ευρώπη. Και εδώ λοιπόν ε, είμαστε στη διαδικασία. Επίσης δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας, τεχνική ομάδα εργασίας μεταξύ των κρατών μελών για ανταλλαγή πληροφοριών για τα ε, κύρια περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την, ε, τις εξορίξεις και επιπλέον η Επιτροπή μελετά τις μελέτες για την χημική ασφάλεια για ορισμένες ενώσεις που χρησιμοποιούνται γενικά για την υδρορογμάτωση για να διευκρινιστεί εάν ε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η έκθεση είναι επαρκής προστασία. Αυτά κάνουμε στον τομέα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τις αρχές, τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα συνεχίσουμε στενά τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Και πάλι το λόγο έχει ο υπογράφων, ο αναφέρον, που είπε ότι θα ήθελε να ε, προχωρήσει σε μια συμπλήρωση της παρέμβασής του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα που τέθηκε. Τι είδους, έχει προσφέ... Τι είδους χρήματα έχει προσφέρει η Σευρών στην ε, βουλγαρική κυβέρνηση. Ξέρετε υπάρχει μια έκφραση ότι άμα θες λεφτά καλύτερα να θες πολλά. Η βουλγαρική κυβέρνηση έκανε έναν διαγωνισμό. Η αρχική τιμή ήταν 250 εκατομμύρια δολάρια. Η Σευρών δήλωσε ότι θα προσφέρει 30 εκατομμύρια δολάρια που θα έπρεπε να επενδυθούν για να αντιμετωπιστούν οι ζημίες στο περιβάλλον. Θέσαμε το ερώτημα αυτό στον πρώην Υπουργό ενέργεια κύριο Τράικοφ, ο οποίος μας απάντησε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν όπως έχει υποσχεθεί η Σευρών στην βουλγαρική κυβέρνηση εφόσον υπογραφεί η σύμβαση. Οπότε τα χρήματα αυτά δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί. Δύο απόψεις κυκλοφορούν κυρίως στη Βουλγαρία οι απόψει των υπέρ και των κατά της ε, εξόριξη του αερίου αυτού. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και βουλγαρικό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι ε, υπάρχει σαφής πλειοψηφία κατά. Διότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται έχει αποδειχθεί σε μια σειρά περιπτώσεις ότι μπορεί να προκαλέσει ζημίες όχι σε όλες. Εξαρτάται βεβαίως από τον, ε, τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. Τι είδους διαστρωμάτωση έχει το έδαφος. Και τώρα έχουν γίνει έγκυρα πειράματα για να αποτιμηθούν οι ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον σε άλλα μέρη. Αλλά στην Βουλγαρία δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και βεβαίω έχω κάθε σεβασμό για τους ε, γεωλόγου της χώρας μου, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη οι απαραίτητε μελέτες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των μελών που πήραν το λόγο το μέλλον αυτής της αναφοράς να παραμείνει ανοιχτά και οι δραστηριότητες της Επιτροπής ε, αποτελούν ένα δίκτυ της προσοχής που πρέπει να αποδοθεί και στο μέλλον και θα ήθελα να προσθέσω ότι διατυπώθηκε και το αίτημα να πραγματοποιηθεί, να διοργανωθεί μια ακρόαση στην Επιτροπή μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει στη συνάντηση των συντονιστών να το συζητήσουμε και μετά από μια βαθύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πάνω στο ίδιο θέμα και για να αποφύγουμε επικαλύψεις εργασιών και για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο λειτουργική την αποτελεσματική την εργασία μας μετά από αυτές τις αναφορές που ακούσαμε Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά και για την ακρόαση που ζήτησαν οι περισσότεροι από τους συναδέλφους θα το αποφασίσουμε αυτό στη συνάντηση των συντονιστών. Να μας μπελιέ που θα ήθελα να έρθει το λόγο στο σημείο αυτό ακριβώς. Μια στιγμή, ναι, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η ακρόαση είναι εντελώς διαφορετική γιατί δεν έχουμε άλλους που έχουν άμεσο ενδιαφέρον από αυτό, αλλά απλά και μόνο μία ακρόαση που αφήνει ακριβώς να συμμετάσχουν ε, οι πολίτες Ευρωπαίοι από τα θέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην περιοχή τους. Είναι κάτι το λοιπόν ε, και όχι ε, πάνω σε αυτό καθ' αυτό. Σόνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή περιβάλλοντος οργάνωσε ήδη κάποιες ε, συνεδριάσεις ε, και ακρόαση για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και την επίπτωσή του ε, στα ύδατα. Και εκεί δεν είχαμε παρά διάφορους επιστήμονες από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και από τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει πάντως μπορούμε να οργανώσουμε ε, και άλλη μία ακρόαση και εκεί θα πρέπει να καλέσουμε περιβαλλοντολόγους ε, έτσι ώστε να είναι παρόντες. Κυρία Κυρία Μπομπίνσκα. Υπήρξε και ακρόαση στην Ήτρε και κάποιες άλλες ακροάσεις. Μπορούν να οργανωθούν και άλλες βέβαια ακροάσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι ποιον ή ποιους θα καλέσουμε διότι έχουμε αναφορά από ε, μια συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά στην ουσία στοχεύει στην απαγόρευση ε, της ε, εκμετάλλευσης ή της εξόριξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και απανταχού της Ευρώπης. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιφέρειες οι οποίες θέλουν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και την εξόρυξή του, γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Επομένως, καλό είναι να γίνει τέτοια, μια τέτοια ακρόαση, αλλά ίσως ε, θα πρέπει ε, να έρθουμε σε επαφή και με την ε, δημόσια, που παίρνουν μέρος στο δημόσιο διάλογο ή, εν πάση περιπτώσει, να καλέσουμε ανθρώπους από διάφορες περιοχές. Πρόεδρο, επί Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις και θα δούμε και τα σχετικά στοιχεία θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών και για το πώς θα οργανωθεί η ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπογράφοντες και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το 17 με δύο αναφορές, την 358 του 2011 του κυρίου Σνάρσκι και 942 2011 Σλόμα Σαντόφσκι 2.200 υπογραφές την πρώτη αναφορά της συνοδεύουν. Και ο κύριος Νάρσκι έχει το λόγο και για τις δύο αναφορές αυτές. Μίσιο. Κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ως νέος Πολωνός, νέος Ευρωπαίος, ήρθα εδώ να υπερασπιστώ τα δικαιώματα πολιτών της Ένωσης. Την αξιοπρέπειά τους, την ταυτότητά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τα άρθρα 2 και 3, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 3, της χάρτας ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα καλούνται τα κράτη-μέλη να σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει όμως να πω ότι η κατάσταση της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Λουθανίας στην Ένωση. Οι Πολωνοί βλέπουν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν την πολωνική μορφή του ονόματό τους να μην γίνεται σεβαστή, καθώς και το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν τα πολωνικά στη δημόσια ζωή τίθεται να αμφιβόλο. Δεν υπάρχει κανένας νόμος ούτω ώστε να υπάρχουν δίγλωσες επιγραφές στη Λιθουανία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να καθορίζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η τελευταία τροποποίηση στον ε, εκπαιδευτικό νομοπλαίσιο κάνει διακρίσεις κατά των πολωνικών σχολείων. Δεν υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι ε, πριν αρχίσουν να ισχύουν αυτοί οι νόμοι. Η Λιουθουανία παραβιάζει βασικές συμβατικές υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η λουθουανική μειονότητα στην Πολωνία απολαμβάνει όλων αυτών των δικαιωμάτων η πολωνική μενότητα στη Λιθουανία πάντα ήταν στην περιοχή αυτή. Οι διακρίσεις αυτές είναι κατά της αξιοπρέπειάς τους, κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους ως πολιτών και κατά της πολυπολιτισμικότητας. Είναι κατά της αρχής της διαφορετικότητας. Αυτής καθε αυτής. Όλα αυτά είναι κατά του άρθρου 4 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία δυσχεραίνεται έτσι η προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Ένωσης. Το γεγονός ότι οι Πολωνοί δεν μπορούν να γράψουν το όνομά τους στη γλώσσα τους δεν είναι συμβατό και με την οδηγία 2043. Οι Λιθουανοί πολίτες ε, πολωνικής προέλευσης δεν είναι αντικείμενο σωστής μεταχείρισης. Είμαι πολίτης της Ένωσης εκτός Λιθουανίας. Αν θέλω να δουλέψω στην ε, Λιθουανία δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την αρχική μορφή του ονόματός μου και φοβάμαι ότι θα υποστώ διακρίσεις λόγω της εθνικότητάς μου. Δηλαδή, το δικαίωμά μου να εργαστώ ελευθέρος παραβιάζεται. Αυτές οι διακρίσεις στη Λιθουανία παραβιάζουν το άρθρο 2 και άρθρο 3 και το άρθρο 4, παράγραφος 3, καθώς και το άρθρο 6 και το άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο 8 και το άρθρο 45 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις ε, διατάξεις οδηγίας 2043. Με συγχωρείτε που μιλάω τόσο γρήγορα. Οι διακρίσει ει βάρο των Πολωνών στη Λιθουανία είναι ασύμβατη με τι γενικέ διατάξει του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα τι ε, ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάζει πολλά άρθρα τη Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 1, το 14, το 15, το 20, το 21 και το 22. Τα προβλήματα που μόλις ε, υπογράμμισα, είναι αρμοδιότητα ενωσιακή. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, διότι είναι παραβίαση αξιών της Ένωσης. Τονίζω επίσης ότι η γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ακριβής και δεν καλύπτει την ουσία του ζητήματος που μόλις περιέγραψα. Η πιο σημαντική πλευρά, δηλαδή η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιθουανία, δεν αναφέρονται καν. Έχει ε, αντιμετωπιστεί με πολύ στενό πνεύμα και έχει διαστραφεί στην ουσία ο τρόπος απάντησης. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία ούτε εγώ δεν ανέφερα και ο τίτλο τη απάντηση νομίζω είναι ανεπαρκή. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση επί τη συνολική επιχειρηματολογία τη αναφορά και θα ήθελα να μου απαντήσει μια πολύ απλή ερώτηση που νομίζω ότι έχει προφανή απάντηση για όλου του πολίτε, Πιστεύει η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή ότι η Λιθουανία, κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να σέβεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Κάθε πολίτη τη Ένωση όπου και αν είναι, όποιοι και αν είναι, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια και να μην παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, νομικά και πολιτικά, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία, ιδιαίτερα τα γλωσσικά τους μειονοτικά δικαιώματα. Οι Πολωνοί που ζουν στην Λιθουανία είναι πολίτες της Ένωσης με πλήρη δικαιώματα και τους αρμόζει κάθε στήριξη και βοήθεια. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση και να επιχειρήσει να διαπιστώσει επιτόπου την κατάσταση. Οι Λιθουανοί και οι, Πολοι, οι Πολωνοί έχουν πολλά κοινά στην ιστορία τους καθώς και στην ιστορία ένταξής τους στην Ένωση. Πιστεύω ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες θα κατορθώσουμε να επιλύσουμε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδι στην αρμονική μας συνεργασία και μέλλον στην Ένωση. Καλό λοιπόν όλους τους ευρωβουλευτές να βοηθήσουν τους Πολωνούς στη Λιθουανία. Αν τους αφήσετε στην τύχη τους, τότε θα αποδείξετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστρέφει τη ματιά από τα προβλήματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι των δύο χωρών, Λιθουανίας και Πολωνίας. Από πλευράς Λιθουανίας, Λίντλα Πελσπλίτελε του Ένε. Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας της Λιθουανίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα, αν μου το επιτρέπετε. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Εξεπλάγημενο από το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς και την κατάθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, εν μέρει διότι το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα δίνει την δυνατότητα στις μειονότητες να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα και εξασφαλίζει την εκπαίδευση στη μητρική τους ε, γλώσσα από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Έχουμε σχολεία λιθουανικά, ε, πολωνικά, ε, λευκορωσικά, τα οποία ε, λειτουργούν στη δική τους γλώσσα στην Λιθουανία. Επομένως, ε, πρέπει να πω ότι δεν ανταποκρίνονται τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην αναφορά ε, στην πραγματικότητα. Γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης ε, και της πολωνικής μειονότητας και δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα, αλλά ούτε προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Η πολωνική μειονότητα στη Λιθουανία έχει δικαίωμα να μάθει την γλώσσα της από το ε, ε, νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο και αυτό αποτελεί μοναδική περίπτωση. Στο Πανεπιστήμιο του Μπιαλιστόκ, στο ε, Βίλνιους, είναι το μόνο τμήμα το οποίο λειτουργεί στα πολωνικά εκτός της Πολωνίας. Πρέπει επίσης να πούμε ότι 10 εκατομμύρια Πολωνοί ζουν εκτός των συνόρων της ε, ε, Πολωνίας και ε, υπάρχουν 70 πολωνικά σχολεία, 55 εκ των οποίων βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μου. Θα πρέπει να πω σαφώς ότι με την ανεξαρτησία της Λετωνίας, της Λιθουανίας, συγγνώμη, ε, αυξήθηκε και ο ρυθμός των πολωνόφωνων σχολείων. Νομίζω ότι με τα στοιχεία αυτά τα μέλη της Επιτροπής θα κατανοήσουν ότι πρέπει πλέον να κλείσουν την αναφορά αυτή. Όμως, ε, και σε σχέση με, τη, με τα στοιχεία, τα εσφαλμένα στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλει οι αναφέροντες, θα ήθελα να υποβάλω στα μέλη της Επιτροπής και κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τροποποίηση του, των εκπαιδευτικών νόμων ε, στην χώρα μου. Άρθρο 30, παράγραφος 1, αναφέρει και παραθέτω ότι τα σχολεία γενικής ε, κατεύθυνσης δημιουργούν προϋποθέσεις έτσι ώστε οι εθνικές μειονότητες να ε, μπορέσουν να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα, να μάθουν την ιστορία τους ε, και την, τον πολιτισμό τους. Τέλος της παράθεσης. Επίσης, ο νόμος ρητά αναφέρει ότι στα σχολεία εθνικών μειονοτήτων ε, ε, γεωγραφία, γεωγραφία, ε, η λιθουανική ιστορία και ο πολιτισμός της Λιθουανίας θα είναι τα μόνα μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται στην λιθουανική γλώσσα. Ε, και ε, αυτό διαφέρει από τον μεγαλύτερο αριθμό των σχολείων απανταχού της Ευρώπης όπου 60% των μαθημάτων ε, διδάσκονται στην χώρα του κράτους στην οποία βρίσκεται το σχολείο. τα μαθήματα στα σχολεία ε, της εθνικής ε, μειονότητας ε, για την Πολωνία, για την περίπτωση της Πολωνίας και της Λευκορωσίας. εκεί έχουμε 90% διδασκαλία στην δική τους γλώσσα και μόνο 10% στη λιθουανική. Επομένως, δίνεται η δυνατότητα ε, να ε, μάθουν τα παιδιά και την δική τους γλώσσα της μειονότητας, αλλά ε, και την λιθουανική γλώσσα, έτσι ώστε να έχουν η εισοδή και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας η διδασκαλία της λιθανικής γλώσσας με κανένα τρόπο δεν διδάσκεται επιζημία της ε, μητρικής πολωνικής γλώσσας ή της ε, γλώσσας της ε, μειονότητας. Ε, η προσπάθεια γίνεται ε, και καταβάλλεται έτσι ώστε ε, οι μειονότητες να εκπαιδεύονται στην χώρα τους. Επίσης, οι κοινοτικές και δημοτικές αρχές έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν μικρά σχολεία γενικής κατεύθυνσης, τα οποία όμως να αφορούν τις μειονότητες ακόμα και με μικρό αριθμό μαθητών, που από 15 έχει πλέον μειωθεί στους 10 η Λιθουανία προετοιμάστηκε σωστά για την εφαρμογή ε, του εκπαιδευτικού νόμου. Όλοι οι καθηγητές που δουλεύουν ε, σε σχολεία της ε, μειονότητας γνωρίζουν καλά την Λιθουανική και αυτό αποδεικνύεται μέσω επιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας και η μεγάλη, η απόλυτη πλειοψηφία των καθηγητών γεωργίας και ιστορίας μετά από την θέση σε ισχύ του νόμου έχουν ε, ε, πάρει και επιπλέον συγκεκριμένα μαθήματα. 800 ε, 800.000 ε, βιβλία και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν μοιραστεί το τελευταίο καιρό στα σχολεία της μειονότητας. Ε, τα εγχειρίδια, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και γεωγραφίας έχουν εκδοθεί ε, σε ειδικές εκδόσεις για τα σχολεία αυτά. Το ζήτημα του, του, της δοκιμασίας, του τεστ ε, για την γνώση της ε, κρατικής ε, γλώσσας έχει ενταχθεί, ε, συγγνώμη, έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταβατικής περίοδου και μάλιστα υπό εξέταση βρίσκεται το ζήτημα της επιμήκυνσης αυτής της μεταβατικής περίοδου. ο ε, πρωθυπουργό Καμπίλα ε, έχει έρθει σε επαφή και συζητά με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον κύριο Τάσκα, έτσι ώστε να συζητηθούν και τα ζητήματα αυτά, καθώς επίσης και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού, του ισχύοντος εκπαιδευτικού νόμου, ε, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υψηλής ποιότητος εκπαίδευση των εθνικών μειονοτήτων. Κατά αυτήν την έννοια την 27η Δεκεμβρίου του 2011 δημιουργήθηκε ε, μία ομάδα εργασίας ε, η οποία εκπροσωπεί όλες τις εθνικές μειονότητες ε, του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο να συζητηθούν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή του εκπαιδευτικού νόμου. νέες πρόνοιες ε, του εκπαιδευτικού αυτού νόμου έχουν ε, συζητηθεί και σε καμία περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο νόμος αυτός ε, προκαλεί διακριτική μεταχείριση. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης της πολιτικής εκδοχής του ονόματος την 12η Μαΐου του 2011 ε, το δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, απεφάνθη ότι οι κανόνες συλλαβισμού και προφοράς των ε, μη λιθουανικών ονομάτων δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε νομική πράξη ή νομικό κείμενο και επομένω, το γεγονό ότι τα ονόματα θα πρέπει να γράφονται με, λιθουανικά, με γράμματα της λιθουανική αλφαβήτου δεν περιορίζει ε, την ελευθερία των ατόμων να χρησιμοποιούν το δικό του όνομα οι εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται και το τονίζω αυτό και το επαναλαμβάνω στην χώρα μας ε, να εκπαιδεύονται λέω στη δική τους γλώσσα από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και αυτό είναι ε, μοναδική περίπτωση καμία οργάνωση, κανένα σώμα δεν απεφάνθη ότι η Λιθουανία παραβιάζει τις υποχρεώσεις της ή τις ενωσιακές αρχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αναφορά αυτή ε, περιέχει εσφαλμένα στοιχεία περί του αντιθέτου ε, και βεβαίω είμαστε στη διάθεσή σα για οποιοδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο Κρίστοφ Τρεβίσκη έχει το λόγο τώρα από πολωνικής πλευράς, σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, διεκριμένα μέλη της Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μου για την δυνατότητα που μου δίνεται να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και την αναφορά που εξετάζουμε. Επίσης, σύντομα θα ασχοληθώ με τα επιχειρήματα της συναδέλφου μου. Χαίρομαι που η διαδικασία αυτή μου θυμίζει την κατά την παράσταση εξέταση στο δικαστήριο, γιατί είμαι δικηγόρος. Πρώτον, ε, είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την απάντηση, ακόμη και της Επιτροπής, σε αυτό το έγγραφο που λέγεται «Σημείωμα προς τα μέλη» της Επιτροπής σας. Όπως ανέφερε ήδη ο, κύριος Αναφέρον, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αναφορά του ήταν ιδιαίτερα στενός ασχολήθηκε μόνο με τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν ασχολήθηκε με τα γλωσσικά αυτά καθεαυτά αιτήματα. Οπότε το κείμενο αυτό δημιουργεί κάποιες συγχύσεις. Δεύτερον, να σχολιάσω τα επιχειρήματα που αναφέρει το σημείωμα της Επιτροπής. Πρώτον, η Επιτροπή αναφέρεται στο άρθρο 165 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό αυτό. Όπου λέγεται ότι τα κράτη-μέλη είναι κυρίως αρμόδια για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και την οργάνωση της εκπαίδευσης με στόχο την ε, διασφάλιση της ε, γλωσσικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας. Στις παρατηρήσεις της ωστόσο, η Επιτροπή αγνοεί τις επιπτώσεις άλλων διατάξεων του Ευρωπαϊκού Νόμου Πρώτον, να θυμηθούμε τι νέα στοιχεία φέρνει το στοιχείο 2 της Συνθήκης για την, για την Ένωση, όπου μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πρόκειται για επαναστατική αλλαγή. Στο παρελθόν, τα αιτήματα σεβασμού των μειονοτήτων αναφέρονταν μόνο στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για υποψήφιες χώρες. Αλλά δεν υπήρχε καμία απέτηση για τα ήδη κράτη-μέλη. Αυτό είχε προκαλέσει επικρίσεις και διορθώθηκε. Γιατί ήταν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έγινε τώρα λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή. Τώρα, οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης εξετάζεται για το εάν και κατά πόσον σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Κάτι άλλο. Θα καλούσαμε την Επιτροπή να επανεξετάσει την άποψή της γιατί έχει και κάποιες άλλες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ας δούμε το άρθρο 10 της συνθήκης. Την άλλη συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης. Εκεί λέγεται ότι κατά τον καθορισμό και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της η Ένωση θα έχει στόχο να καταπολεμήσει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλλο, τον φιλετικό, εθνοτικό κλπ. Ε, λόγο. Αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι παίρνει πολύ ενεργητική, υιοθετεί πολύ ενεργητική στάση όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων, όχι την παθητική στάση που είχαν προηγούμενες διατάξεις αλλά βεβαίω και στο άρθρο 6 υπάρχουν μερικές ε, συμπληρωματικέ ε, δυνατότητε. Η Επιτροπή στην παράγραφο 3, σελίδα 2 του κειμένου της, αναφέρεται σε επιχειρήματα που αφορούν το άρθρο 21 και 22 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και βεβαίως, σωστό αυτό. Αμέσως ευθύς εξ αρχής αναφέρεται και στο άρθρο 51 που θέτει το συγκεκριμένο πλαίσιο για την εφαρμογή της ε, χάρτας αναφέροντας ότι επειδή η χάρτα αφορά τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη και τονίζει ότι δεσμεύονται από την συνθήκη αυτή όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Όμως, Οι διατάξεις καταπολέμησης ε, των διακρίσεων των διαφόρων αυτών κειμένων αγνοούνται. Ας πάμε στην ε, Οδηγία 2043. Αναφέρεται εκπεφρασμένα η εκπαίδευση ως τομέα, όπου πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ε, για την, τις μη διακρίσεις. Επίσης, Αναφέρομαι στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της συνθήκης Λισαβόνας που λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών θα αποτελέσουν τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου. Γενικές αρχές. Θα διευκόλυνε αυτό το μέσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει καλύτερα τα αιτήματα αυτά. Τώρα, λίγα λόγια ε, σε αυτά που είπε η συνάδελφός μου. Έθιξε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκαν από τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις για τα θέματα εκπαίδευσης. Βεβαίως, συστάθηκε μια τέτοια ομάδα εργασίας, συνεδρίασε πέντε φορές και στην πέμπτη τελευταία συνεδρίασή της δεν δημοσίευσε καμία έκθεση ή καμία σύσταση. Ενδιαφέρον. Δεν νομίζετε. Έγιναν συζητήσεις, αλλά δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα. Η λιθουανική άποψη, κατά τη γνώμη μας, δεν συμφώνησε σε καμία τροποποίηση του νόμου για την εκπαίδευση. Πρόκειται για ομάδα εργασία μεταξύ των δύο κρατών. Και αυτό ήταν ε, οπωσδήποτε απόρρια των διακρίσεων που υφίστανται. Δεν θα πέρασω τώρα στον τρόπο γραφή των ονομάτων. Χαίρομαι που η συνάδελφός μου δεν έχει κανένα πρόβλημα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης Πλαίσιο. Κάθε φορά που υπήρξε ε, έκθεση από πλευρά Λιθουανία υπήρξαν επικρίσει. Και μάλιστα η Λιθουανία υποσχέθηκε να τροποποιήσει τον νόμο, αλλά δεν τήρησε την υπόσχεσή τη. Σα παρακαλώ να λάβετε υπόψη όλα τα επιχείρηματα αυτά. Στηρίζουμε λοιπόν τι προτάσει του αναφέροντο να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα έκθεση που να αντιμετωπίζει με πιο ανοιχτό πνεύμα και λιγότερη αλλεργία. Αντιλισαβονική αλλεργία, τα θέματα αυτά θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε και εμείς να σε ευχαριστήσαμε για αυτή την εισήγησή σας με πολλές λεπτομέρειες. εκπρόσωπος της Επιτροπής τώρα έχει το λόγο. Αντώνιου Μάρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει γραπτή απάντηση για την αναφορά αυτή, για τον τρόπο με τον οποίο υπευλήθη αρχικός καθώς επίσης ε, και ε, στη σχέση με την ε, συμμόρφωση προς, τον Ευρωπαϊκό, προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έτσι όπως αναφέρεται στο άρθρο 213 της Συνθήκης Λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ζήτημα το οποίο υποβάλλεται από τον αναφέροντα, δεν εμπίπτει σε τις αρμοδιότητες, γιατί ε, το άρθρο το οποίο ανέφερα προηγουμένως ρητά αναφέρει ότι το κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο αποφασίζει για την γλωσσική του στρατηγική, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό του σύστημα. Επίσης, όλες ε, οι πρόνοιες ε, και οι διατάξεις οι οποίες αναφέρθηκαν από τον αναφέροντα, δηλαδή ε, συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των ε, μειονοτήτων, ε, συνθήκη για το θεμελιώδη, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ. δεν εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν δικαιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί σε παραβιάσεις των εν λόγω διεθνών κειμένων. Όσον αφορά την ίδια τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις διατάξεις της, Αυτές οι διατάξεις ε, απευθύνονται μονάχα στα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν και υλοποιούν ε, το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Σύστημα. Μονάχα σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει την επιβολή της συμμόρφωσης. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται εδώ είναι νέα, διότι δεν είχαν αναφερθεί στην αρχική αναφορά. Τα άρθρα 2, 3 ή 10 4 ή 10, καθώς επίσης και οι διατάξεις τις οδηγίες 243 που αφορούν ε, την διακριτική μεταχείριση βάσει της εθνότητας ή της γλώσσας. Δεν θα έχουμε χρόνο να απαντήσουμε νομίζω σε κάθε ένα από τα επιχειρήματα εν λεπτομερία γιατί κάτι τέτοιο θα προαπαιτούσε νομική ε, ανάλυση, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει ε, την τελευταία στιγμή και με βιασύνη. Μπορώ όμως να σας δώσω μια κατεύθυνση ε, σε σχέση με το πού θα εστιάσουμε την ε, ε, απόφασή μας, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Ας πούμε το άρθρο 10, το οποίο ρητός αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, the Union shall, και επομένως εδώ αναφερόμαστε σε παραβίαση από πλευράς των κρατών την οδηγία 200 2000 ε, πρέπει να σας πω ότι εδώ μιλάμε, ε, ε, εδώ γίνεται λόγος για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ εσείς αναφέρεστε στο περιεχόμενο της, του εκπαιδευτικού συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε πάλι εκτός του πεδίου εφαρμογής. μέσα στο στενό πλαίσιο της δικιάς μας αποστολής, της επιβολής δηλαδή συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της συνθήκης, εδώ ε, είναι σαφές ότι τα αναφερόμενα ε, δεν εμπίπτουν εις ε, την δικαιοδοσία της επιβολής. Είναι εκτός πεδίου εφαρμογής λοιπόν της δικιάς μας επιβολής συμμόρφωσης. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον Βαλέσα. Ευχαριστώ. Η αναφορά του κύριου Σμάρσκι ε, θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης της πολωνικής μειονότητας και της πολωνικής γλώσσας στη Λιθουανία. στο εμπαρόδο η πολωνική μειονότητα είναι η μεγαλύτερη στην χώρα αυτή δεν υπάρχουν αρκετά σχολεία ε, με πολωνική γλώσσα. Ε, δεν μπορούν οι Πολωνοί ε, να προφέρουν τα ονόματά τους με, τον Πολωνί, με την πολωνική προφορά. Η ρύθμιση σχετικά δεν μπορεί έτσι να αφαιθεί στα χέρια των κρατών μελών, γιατί παρόμοιες ενέργειες οδηγούν στην εγκατάλειψη του σεβασμού των θεμελιωδικών δικαιωμάτων στα οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελεύθερη διακίνηση ε, των πολιτών και η ελεύθερη έκφραση στη γλώσσα τους. Αυτά όλα έχουν μεγάλη σημασία για κάτι το εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς προσωπικά υποστηρίζω την αναφορά και θα ζητήσω από αδέλφους να κάνουν το ίδιο. Για τον κύριο Σνάρχη να συμπληρώσω κάτι. Εσείς ε, είστε, είσαστε στην Λιθουανία και διαπιστώσατε τα προβλήματα τα, εκεί τα προβλήματα των Πολωνών στη Λιθουανία. Έχετε υποστεί ο ίδιος ε, διακρίσεις επειδή είσαστε Πολωνός εκεί και τι γίνεται ακριβώς με αυτές ε, με, με τις μειονότητες Κασούμπα ή την ε, λιθουανική μειονότητα στην Πολωνία και υπάρχει παραβίαση τέλος πάντων αυτών των δικαιωμάτων εκεί και τι προσδοκίες έχετε σε σχέση με την αναφορά σας. Ευχαριστώ ο ο κύριος Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω το περιεχόμενο της αναφοράς του κυρίου Σμάρσκι. Αναφέρεται σε συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος μέλος, το οποίο κατηγορείται ότι περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ατόμων. Πολλές ανοησίες βλέπω εδώ, τα οποία δεν χρειάζονται ούτε να τα σχολιάσει κανείς. Αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι ότι όχι μόνο η Λιθουανία είναι κακή, ίσως η χειρότερη από τις γειτονικέ χώρες, από την ε, Ρωσία μέχρι την ε, Γερμανία, αλλά και η Κομισιόν είναι κακιά και αυτό είναι κάτι καινούριο. Βλέπω εδώ τώρα το σημείωμα προς τα μέλη. Πολλές ε, ε, κατηγορίες Κανείς ε, δεν δέχεται ότι κατηγορείται η Λιθουανία. Βλέπουμε εδώ ότι κατηγορείται η Λιθουανία γενικώ για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση κτλ. Φαίνεται ότι τα ξέρει πολύ καλά αυτό ο αναφέρον και αναφέρεται στο, δεν αναφέρεται μόνο στο, στην στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πολωνική μειονότητα με την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα με τον τρόπο που η Λιθουανία αντιμετωπίζει τις ε, μειονότητες ε, της Πολωνίας, της Λευκορωσίας. Ε. Ίσως ε, και οι τελευταίες μη φιλικές κινήσεις ε, και αποφάσεις ε, του Πολωνικού Υπουργού Εξωτερικών να έπαιξαν κάποιο ρόλο. Αναφέρεται επίσης ότι τα μέλη της μειονότητας της Πολωνίας δεν, δεν έχουν το δικαίωμα να εκπαιδευτούν στην γλώσσα τους όταν ζουν στην Λιθουανία. Βεβαίως, μέσα σε δύο χρόνια τα, η γεωγραφία, ας πούμε, ή η ιστορία ε, αναφέρεται ότι θα πρέπει να διδάσκονται ε, στην ε, κρατική γλώσσα σε δύο χρόνια δεν ξέρω, ίσως να μην έχουν μάθει μέσα στα μέχρι 20 χρονών, να μην έχουν μάθει καν τη λιθουανική γλώσσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην μπορούν δηλαδή ούτε καν αυτά τα μαθήματα να διδαχτούν στην χώρα αυτή. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν μπορεί να συσταλεί ε, το δικαίωμα ε, να γνωρίσουν τα γεωγραφικά ονόματα στην, ε, χώρα, στο κράτος, στο, κράτος αναφοράς. Φαίνεται ότι δεν συμφωνεί ούτε με αυτό η αναφορά. Και μετά ακολουθεί και η σύνοψη της αναφοράς. Λέμε, αναφέρεται ότι η κρατική γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την διδασκαλία της ιστορίας και ε, της ε, γεωγραφίας ε, συμπεριλαμβανομένων και των πολωνικών σχολείων. δεν καταλαβαίνω εγώ τι γίνεται εδώ. Γιατί η διδασκαλία της γεωγραφίας δημιουργεί πρόβλημα. Ε, και καταλήγει αναφορά στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι ε, η διδασκαλία στην κρατική γλώσσα των δύο αυτών μαθημάτων μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ε, να μειώσει τον αριθμό των μαθητών και επομένως να κλείσουν τα σχολεία. Η μείωση των η μείωση των μαθητών στα σχολεία είναι μάλλον αποτέλεσμα ε, του ελληπούς βαθμού αγάπης μεταξύ των συζύγων, θα έλεγα εγώ. Και βεβαίως μπορεί να είναι ατυχής αυτή η κατάσταση αλλά, και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των μαθητών. Γι' αυτό κλείνουν τα σχολεία. Αλλά και στην Πολωνία κλείνουν τα λιθουανικά σχολεία. Ε, λόγω του ε, μειωμένου αριθμού μαθητών όπως ε, αναφέρεται. Αλλά η μείωση των αριθμ, του αριθμού των μαθητών δεν εξαρτάται από τη διδασκαλία της ιστορίας της γεωγραφίας σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν γίνεται η διδασκαλία αυτή. Καλό λοιπόν τον κύριο Σνάσκι που υπέγραψε αυτήν την αναφορά να του πω ότι αυτό το κείμενο το οποίο υπέγραψα δεν είναι σοβαρό. Ε, γίνεται αναφορά ε, στη υποτιθέμενη μείωση των, ε, της διδασκαλίας των πολωνικών και, βάση περιπτώσει, τι να σας πω, εγώ δυστυχώς τα διαβάζω όλα αυτά, νόημα πολύ δεν βγάζω, και γι' αυτό σας παρακαλώ μην μας παταλάτε το χρόνο μας με τέτοια ζητήματα. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίζουν να λένε τα ίδια και τα ίδια. Ε, τα έχουμε ξανακούσει Αυτέ Αυτά, αυτές ε, ε, ε, έχουν γίνει δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα τραβήξουν το αυτή της Λιθουανίας και η Ευρωκομισιόν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Και τελικά δεν φτάνουμε σε κανένα συμπέρασμα. Δεν δίνονται νέα στοιχεία, δεν εξάγονται νέα συμπεράσματα. Και φαίνεται ότι είναι, τελούν συγχύση οι ίδιοι και προκαλούν σύγχυση και σε όλους και σε, όλα τα, ε, σε όλες τις βαθμίδες της ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας. As well. Thank you. Thomas... Ε, κύριε Στομασέσκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Πολύ δύσκολο να σχολιάσω αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον ε, προηγούμενο μιλητή. Αλλά δεν είναι πολύ σοβαρή αντιμετώπιση. Ένα μέλος της Επιτροπής μας να αντιμετωπίζει έτσι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πραγματικό, πρέπει να τονίσω, και δεν αφορά μόνο την ε, εκπαίδευση των ε, εθνικών ε, μειονοτήτων. Εγώ, ως Ευρωβουλευτής, αναγνωρίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και αυξήθηκαν τα προβλήματα αυτά μετά την ένταξή μας στην Ένωση. Είναι παράδοξο βεβαίως αυτό. Οι εθνικές μειονότητες συμμετείχαν ενθουσιαστικά στο δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ένωση. Πολύ ψηλή συμμετοχή, πολύ ψηλό ποσοστό υπέρ της Ένωσης και μόλις ε, γίναμε μέλος της Ένωσης ε, άρχισαν τα προβλήματα και όχι μόνο στον τομέα της ε, εκπαίδευσης. Το 2009 καταργήθηκε από το Κοινοβούλιο ο νόμος για τις εθνικές μειονότητες. Είμαστε μάλλον η μόνη χώρα όπου δεν υπάρχει νόμος για τις εθνικές μειονότητες νόμος που είχε εγκριθεί το 1991 μόλις η χώρα μου ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Ανεξαρτησία για την οποία παλέψαμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Είμαστε στο δρόμο διαμαρτυρώμενοι κατά του καθεστώτος και καταφέραμε να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας. Οι Πολωνοί και οι άλλες μειονότητες υποστήριξαν την ανεξαρτησία της Λιθουανίας και μετά τα αιματηρά γεγονότα του Ιανουαρίου ψηφίστηκε αυτός ο θαυμάσιος νόμος για τις εθνικές μειονότητες τον οποίο υπέγραψε ο συνάδελφος κ. Λαντσμπέργης που ήταν τότε πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου και το ίδιο λοιπόν πολιτικό κόμμα στο οποίο πάντα ανήκει ο κ. Λαντσμπέργης δυστυχώς το 2009 μετά την ένταξή μας στην Ένωση κατήργησε αυτό το νόμο τώρα πια δεν έχουμε τα δικαιώματα για τα οποία αγωνιστήκαμε με τόσο πάθος. Ένα τμήμα λοιπόν του λαού μας έχει δυσχέρειες. Εάν χρησιμοποιήσει την μητρική του γλώσσα στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να πληρώσει πρόστιμα, όχι μόνο για δίγλωσες επιγραφές. Στους δρόμους αλλά ακόμη και αν υπάρχει ε, μία επιγραφή σε ένα λεωφορείο, σε ένα κατάστημα. Σύμφωνα με τον νόμο, που όπως σας είπα καταργήθηκε το 2009, οι εθνικές μειονότητες σε ορισμένες περιοχές, για τις ορισμένες περιοχές οι εθνικές μειονότητες 80% του πληθυσμού. Φανταστείτε λοιπόν την κατάσταση. Υπάρχουν 14 δήμοι, σε, μερικές, σε μερικούς από τους οποίους 80% του πληθυσμού είναι εθνικές μειονότητες. Και δεν έχουν δικαίωμα ο δρόμος να αναφέρεται στη γλώσσα τους. Οι πινακίδες για τους δρόμους. Και αν κάποιος το κάνει, αν κάποιος λοιπόν στη δημόσια σφαίρα χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, μπορεί να πληρώσει έως και 500 λίτας για τη χρήση της, μητρική τους, της μητρικής τους γλώσσας στις περιοχές όπου, ξαναλέω, 80% του πληθυσμού είναι τμήμα της πολωνικής μειονότητας. Αυτό προκύπτει επίσης ε, στον τρόπο γραφής των ονομάτων και επωνύμων. Δεν είναι δυνατόν να εμποδίσουν τους ανθρώπους να γράψουν το όνομά τους όπως θέλουν. Όταν ήμουν 16, το 1981 στη Σοβιετική περίοδο αρνήθηκα να πάρω Σοβιετικό διαβατήριο και τότε με επισκέφθηκε η Σοβιετική πολιτοφυλακή και μου είπε δεν μπορείτε να υπάρχετε νομοθετικά χωρίς διαβατήριο ή ταυτότητα. Και τους είπα δεν το θέλω γιατί δεν γραφετε σωστά το όνομά μου σε αυτό το έγγραφο. Και ενώ ήταν τότε απολυταρχικό το καθεστώς, ολοκληρωτικό, δέχτηκαν να γράψω το όνομά μου στη μητρική μου γλώσσα και τώρα δεν το δέχονται. Φυσικά δεν είναι ικανοποιημένη η πολεμική μειονότητα με την κατάσταση αυτή. Στις 17 Μαρτίου μάλιστα υπήρξε μια διαδήλωση με συμμετοχή περίπου 10.000 ατόμων. Βγήκαν στους δρόμους. Μέλη του Συνδικάτου των ε, Δασκάλων και Καθηγητών αλλά και άλλοι. Τονίζω λοιπόν ότι η αναφορά αυτή δεν είναι κατά της Λιθουανία, είναι κατά της ε, κυρίαρχης πλειοψηφία, της κυβερνώσεω ε, πλειοψηφία, γιατί και η αντιπολίτευση, οι σοδημοκράτε κατακρίνουν αυτόν τον νόμο. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε. Διαφορετικά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τι εργασίες μα και άλλοι πολίτε θα πρέπει να λάβουν το λόγο. Γι' αυτό Σα παρακαλώ σύντομα. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο πάλι. Θα είμαι σύντομη. Εάν ισχυρισμοί... Κοιτάξτε, ακούμε αντικρουόμενα επιχειρήματα. Αλλά πρώτον να πω προς την Επιτροπή ότι ακόμη και αν δεν μπορούν να κάνουν προσφυγή κατά της Λιθουανίας έχουμε κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Δεύτερον, δεν θα μπορούσατε να στραφείτε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί είναι θέμα αρμοδιότητάς του. Πρόκειται για το δικαστήριο στο Στρασβούργο. Και κάτι τελευταίο. Επανειλημμένα έχουμε απασχοληθεί και με την ρωσική μειονότητα στις βαλτικές χώρες, που έχει ακόμη χειρότερα προβλήματα τους στερούν θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορούμε λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και θα πρέπει. Αλλά θα υπάρχουν κάποιοι που να μπορούν να μας πούνε ποια είναι η πραγματικότητα. Λεγκούτκο. Κοιτάξτε, το θέμα είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, ένα σύντομο σημείο το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Κοιτάξτε, ας κάνουμε ένα ε, πνευματικό πείραμα, θεωρητικό πείραμα. Ας πούμε ότι είστε ξαφνικά σε μια χώρα στην οποία μια ωραία μέρα το όνομά σας που έχετε χρησιμοποιήσει για πολλά χρόνια που ήταν το όνομα του πατέρα σας, του παππού σας μια μέρα λοιπόν δεν έχετε πλέον δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα. Είστε κάποιο άλλο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ε, Σα ευχαριστούμε, συνάδελφε. Βάλεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αφενός είναι προφανές για όλους μας ότι η κάθε χώρα μας βάσει εθνικού σχεδίου ε, οργανώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά μπορεί να αντικαταστήσουμε τη Λιθουανία από μια άλλη χώρα και την πολιτική μειονότητα με μια άλλη μειονότητα και το πρόβλημα ξαναρχίζει και είναι το ίδιο. Σε ποια γλώσσα διδάσκεται η γεωγραφία και η ιστορία. Επίσης συνεχίζεται μετά στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υπάρχει η, επίσημη γλώσσα της χώρας ή η, χώρα, η γλωσσα της μειονότητας. Αυτά δεν είναι εξειδικευμένα προβλήματα. Είναι ε, κοινά σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν μειονότητες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν ε, ασκήσουμε κριτική σε οποιαδήποτε κατάσταση χωρίς να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά περιστατικά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια συγκινησιακή φόρτιση πάντα όταν συζητούμε ε, τα θέματα αυτά. Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στην ίδια Ήπειρο. Θα πρέπει λοιπόν ε, με ηρεμία και χωρίς θυμικές εξάρσεις να δούμε κατά πόσον εφαρμόζεται ο νόμος και αν εφαρμόζονται και οι ενωσιακές διατάξεις για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Καλνόσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την εφαρμογή αυτού του νέου Μητρώου στη Λιθουανία αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, αλλά ποιο είναι το βασικό πρόβλημα το πώς θα έχουμε μία ενιαίες εξετάσεις, ενιαίο τεστ σε όλα τα σχολεία και στα σχολεία των μειονοτήτων. Ε, το, η τελική εξέταση θα πρέπει να είναι η ίδια όπως και στα λιθονικά σχολεία. Στα σχολεία των μειονοτήτων υπήρχε μια τελική εξέταση στη γλώσσα της χώρας, αλλά είχε να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο το πραγματοποιούσαμε μετά από 12 χρόνια εκπαίδευσης ε, και ήταν ακριβώς ένας εξετάσεις κάπως ε, χαμηλότερο επίπεδο. Τώρα εδώ επιτρέπεται σε τρία, ε, μάλλον σε τρία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία εξέταση και αυτό δεν είναι σωστό εδώ. Είναι, γίνεται διάκριση γιατί εδώ αφορά μόνο τρία χρόνια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί γιατί είναι δικαίωμα του λιθανικού κράτους γενικά, αλλά αυτή η διάκριση όμως είναι σκανδαλώδης. Και ακόμα ασχολήθηκα με το θέμα και για τη ε, μειονότητα στη μία χώρα και στην άλλη όταν ήμουν ακόμα μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου. Και είχα συλλογιστεί πολλά και διάφραγματα για όλα αυτά τα επιχειρήματα που δόθηκαν για να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ είχαμε διάφορες μελέτες κοινωνιολογικές με διάφορες ερωτήσεις ε, στα μέλη των μειονοτήτων και τους ζητούσαν ε, ανάμεσα στις ερωτήσεις να απαντήσουν. Θεωρείτε ότι μια ελλειπής γνώση της εθνικής γλώσσας ε, μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για το εξέβεση εργασίας και το 30% είχε πει ναι, αν δεν γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα της χώρας μπορούσαμε να έχουμε εμπόδια για να αναζητήσουμε εργασία. Αλλά τα ίδια αυτά άτομα όταν ρωτήθηκαν εσείς αντιμετωπίσατε δυσκολίες να βρείτε δουλειά επειδή είχατε δυσκολίες στη γλώσσα της χώρας μόνο το 3% απάντησε ναι αλλά από την κοινωνιολογική έρευνα είχε αναφερθεί μόνο η πρώτη απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή δεν έχει τις σωστές πληροφορίες γιατί λένε το 30% του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες να βρει δουλειά επειδή δεν ξέρει την εθνική γλώσσα γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Αλλά είναι, είναι αλήθεια, είναι μόνο το 3% που έχει το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Λιθουανία θεωρεί ότι οι μειονότητες είναι άρρηκτο τμήμα της πολιτιστικής της κληρονομιάς ε, και της εθνικής της υπόστασης έχουν ε, υπάρξει εξαιρετικές ε, υποδειγματικές συνθήκες εκπαίδευσης για την πολωνική μειονότητα. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Λιθουανία αφορά ε, την βελτίωση συνθήκων για όλους τους μαθητές, ε, ανεξαρτήτως του αν ανήκουν σε κάποια μειονότητα ή όχι. Η Λιθουανία είναι η μοναδική χώρα η οποία δίνει την δυνατότητα σε Πολωνούς ε, να εκπαιδεύονται από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής τους διαδρομής στην Πολωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ε, είναι καλύτερο ε, να ε, γνωρίζει κανείς καλά και την γλώσσα του κράτους το οποίο ζει. Ο κύριος Κορονόφσκι είπε προηγουμένως ότι δεν είχαν πρόβλημα οι Πολωνοί της Λιθουανίας να βρουν δουλειά εάν δεν ήξεραν τα, πολωνικά, τα λιθουανικά και επομένως γιατί φοβούνται να υποστούν αυτό αυτή την γλωσσική δοκιμασία. Ο κύριος Τομασεύσκη ανέφερε προηγουμένως ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα ε, ε, και ότι είναι κατά της ε, λιθουανικής κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως και μια ομάδα εργασίας διακρατική και αναφέρθηκε ότι η λιθουανική πλευρά μαζί με την πολωνική αποφάσισε ε, η μεταβατική περίοδος να μην είναι διετής αλλά οκταετής. Δεν ξέρω γιατί δεν υπεγράφει τελικά αυτό. Ο Υπουργός... Ε, ε ο Υπουργός ε, εκπαίδευση της Λιθουανίας είπε στον ΙΠΑ το εκπρόσωπο για του ΟΑΣΕ για θέματα εκπαίδευση ότι βεβαίω ε, η λιθουανική γλώσσα θα πρέπει να, γίνει, να, να είναι γνωστή αλλά από την άλλη πλευρά ε, η μεταβατική περίοδος θα, θα κρατήσει, θα διατηρηθεί μέχρι ότου αυτοί που έχουν ξεκινήσει στη μειονοτική εκπαίδευση να ολοκληρώσουν το σχολείο. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται μία προσπάθεια να ε, πείτε τα πράγματα με το όνομά, με τους όσον αφορά την ιστορία και τη γεωγραφία. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω εγώ σε όσα, για όσα είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ήταν η κλασική στάση νομική απέναντι σε παρόμοια προβλήματα. Η κατάσταση αυτή δεν είναι κάτι το καινούριο. Εδώ και αρκετά χρόνια οι Πολωνοί στη Λεθωανία παραπονιούνται για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και αναφέρουν περιπτώσεις διάσκηση διάκριση. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει σαν ρόλο να συμφιλιώνει τις δύο πλευρές και να μειώνει τι διαφορέ του και να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητού. Δεν θα έπρεπε να κάνει αναφορές μόνο σε νομικές ρυθμίσεις, άρθρα κλπ. Εδώ το σχέδιο ευρωπαϊκής οικοδόμησης είχε σαν σκοπό να εγγυηθεί μια ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα έλυναν τα προβλήματά τους και θα αποφεύγαν τις σειράξεις. Σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, γιατί υπήρχε στη σύσταση του φορέα της εταιρείας για τα ανθρώπινα, του Ιδρύματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει το τι θα γίνει. Θα χρειάζεται να δούμε τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και να μπορέσουμε μετά να παρουσιάσουμε μια έκθεση και να κάνουμε μια εκτίμηση που ίσως ε, για τη μία ή την άλλη πλευρά και τις δύο να μην ήταν και τόσο άνετη και καλή. Αλλά αυτό το Ινστιτούτο, γιατί εμείς προχωρήσαμε στη σύστασή του, θα ζητάω από την Πρόεδρο να εξ ονόματος της Επιτροπής να προσκαλέσει και αυτό το φορέα. Ο κ. Μποστινάρου τελευταίος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, φρονώ πως ε, το θέμα είναι ιδιαίτερα συγκινησιακό. Ε, είναι ευαίσθητο ζήτημα γιατί αφορά την ταυτότητα και τις ταυτότητες και μερικές φορές ε, υπάρχει σύγκρουση ταυτοτήτων ε, που μπορεί να καταλήξει σε ανοιχτές σειράξεις όπως το έχουμε δει στο παρελθόν στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ευαίσθητο και συγκινησιακό. Πιστεύω λοιπόν ότι το μόνο που μπορεί να κάνει η Επιτροπή μας είναι να συζητήσει το ζήτημα όταν θα έχει πρώτερη αξιολόγηση. Η μόνη αξιολόγηση την οποία θα μπορούσα να σκεφτώ είναι αυτή ε, του είπα του εκπρόσωπου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων του ΟΣΕ, καθώς επίσης και την αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για την εφαρμογή των, ε, της Χάρτας των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων στις ε, εν λόγω χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την δυνατότητα και δεν είναι προετοιμασμένη να κάνει αξιολογήσεις όσον αφορά τα γλωσσικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων κτλ. Είχαμε ένα αντίστοιχο ζήτημα όταν συζητούσαμε το Ουγγρικό Σύνταγμα και τον ε, Ουγγρικό Νόμο για τα μέσα ενημέρωσης ε, και το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΕΣΕ ε, είπαμε ότι θα πρέπει να αποφανθούν. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε αξιολόγηση της κατάστασης από αυτά τα δύο όργανα για να δούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα δικαστεί, θα εκδικαστεί η υπόθεση ή να αποφανθούμε μέσω τιμιγορίας υπέρ του ενός ή του άλλου από την εμπειρία μου ως Ρουμάνου, όπου η έλλειψη δικαιωμάτων ε, των μειονοτήτων μπορεί να οδηγεί, μπορεί να οδηγήσει ε, σε περιπλοκές, ενώ η υπερβολική αύξηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων μπορεί ε, να οξύνει προβλήματα. Κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Καλό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εσάς να δείτε με ποιο τρόπο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, έτσι ώστε να ζητήσουμε από αυτά τα δύο όργανα μία αξιολόγηση της νομικής κατάστασης, ε, της ε, εφαρμογής των νόμων να αποφανθεί εάν ναι ή όχι υπάρχουν παραβιάσεις ή διαπιστώνονται παραβιάσεις ε, στην ε, εφαρμογή του νόμου και τότε η Επιτροπή ε, να πάρει την απόφασή της έχοντας στα χέρια της τις δύο αξιολογήσεις μα είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν ότι είναι θέμα επικουρικότητα. το κράτο μέλο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει. Ε, το ξέρουμε όλο αυτό το, την ιστορία σχετικά με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κτλ. Η κατάσταση είναι ευρύτερη. Εάν δει κανείς τις χώρες της Βαλτικής, κατανοεί ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με χώρες, ε, υπάρχουν προβλήματα με μειονότητες, υπάρχουν προβλήματα με απάτριδες, υπάρχουν προβλήματα με ανθρώπους ε, στους οποίους αρνούμαστε την έκδοση διαβατηρίου και στο όνομα των αρχών ε, το, τις οποίες ε, προασπίζουμε πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από λογική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ στην Μπροστινάρου. Θα ξαναδώσω το λόγο στον ε, αναφέροντα για δύο λεπτά έτσι ώστε να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο, δύσκολο είναι σε δύο λεπτά να απαντήσω σε ό,τι υπόθηκε αλλά εδώ έχω δύο έγγραφα την αναφορά μου και μετά από δίπλα το κείμενο της Επιτροπής. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρατε ότι εξαιτία του περιορισμού της διδακτέας ύλη μειώθηκε ο ρυθμός των σχολείων αλλά μειώνεται όμως ε, ο αριθμός των σχολείων. Εδώ στην αναφορά μιλάμε πολλές φορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ δεν εμφανίζεται πουθενά στο κείμενο της Επιτροπής αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης υπάρχει και ένα παράρτημα στην αναφορά μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα εκπαίδευσης, μόρφωσης. Ε, κύριε Λαντσπέργης, εγώ ιδιαίτερα σας σέβομαι για όλα όσα κάνατε για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί πρόβλημα και πολεμική με την κυβέρνηση. Εδώ δεν είναι θέμα κυβέρνησης, αλλά είναι η φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητάνε βοήθεια και μια, μια ένδειξη αλληλεγγύης. Αυτά και ε, ε, ακούστηκαν κριτικές ε, για πράγματα που εγώ δεν έχω γράψει καθόλου. Βλέπετε εδώ όλη την αλληλογραφία με την γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Είπα ότι υπήρξαν και διάφορα που δεν στέκουν ψεύδι και τα πράγματα όμως τα πήραν ιδιαίτερα στα ελαφρά. Παρακαλώ να επανεξετάσετε την αναφορά μου με όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησα. Σας ευχαριστώ επίσης για την υποστήριξή σας. Και εδώ να σας πω ότι τα μέσα ενημέρωση στη Λιθουανία όταν αναφέρθηκαν στην αναφορά μου έγραψαν το όνομα και της Επιτροπής Αναφοράς λάθος. Εσείς δεν το βλέπετε όμως εδώ πέρα. Και Ε, επισκέπτομαι ας πούμε με ένα νεκροταφείο στη Ρωσία και τι βλέπω ότι η Πολωνοί δεν αντιμετωπίζουν με δύο τρόπο. Ε, η Λιθουανία μπορεί να είναι ένα υπέροχο αριστό μέλος. Ελπίζω να υπάρξει μια υπάρξει μια συνεργασία. Το ίδιο και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δυστυχώ κάτι που δεν συμβαίνει. Και ήμουν σε επαφή και με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Το Ίδρυμα που υποστηρίζει τους Πολωνούς στο εξωτερικό, πολίτες στο εξωτερικό. Και επίσης με δύο μη κυβερνικές οργανώσεις στη Λιθουανία. Και από τις εκθέσεις τους ε, ε, επιβεβαιώνονται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιθουανία. Το 1967 ακούσαμε μια κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που έλεγε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέρος του κοινοτικού και εκτιμένου. Στο Τζάντσιχ είμαι ε, φοιτητή εγώ και όλοι γνωρίζουν ότι είναι από τις βασικές αξίες τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω κάτι ότι η αναφορά μου ουσιαστικά αποτελεί τη φωνή, το αίτημα για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κατάλληλες ενέργειες που θα εγγυηθούν την ισότητα, τα ίδια δικαιώματα για όλους. Από την Επιτροπή σας, ο κ. Βέντσα είπε τι περιμένω εγώ, τι προσδοκώ. Θα ήθελα να παροτρεθούν όλα τα κρατημέρη να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η Επιτροπή δεν απάντησε στο ερώτημά μου. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν χρέος να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι ή όχι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετέ φορέ υιοθέτησε παρόμοια ψηφίσματα ψηφίσματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σχετικά με την Πολωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2012, ναι, θα θέλω να πω ότι η γερμανική γλώσσα, ας πούμε, σε 33 δήμους υιοθετήθηκε στην Πολωνία σαν δεύτερη γλώσσα. Και το ίδιο είναι και στις δύο γλώσσες, ρωσικά κλπ. Και θα ήθελα όμως ε, να ακούσω μια συγκεκριμένη άποψη. Εδώ το ζητάω σαν πολίτης και όχι σαν ε, κυβέρνηση της Λευθανίας Ευχαριστώ. Θα κάνω μια εξαίρεση. Ο Στένφος Κάσμαν που έφτασε μόλις τώρα θα ήθελα να κάνω μια εξαίρεση να του δώσουμε για ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να είμαι στην άλλη επιτροπή για ε, την οποία είμαι μέλος ε, γιατί έπρεπε να ψηφίσουμε. Όμως να στηρίξω την αναφορά αυτή. Υποστηρίζω αυτά που μόλις ε, ακούστηκαν από πλευρά από ε, ε, προοπτική ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μπορώ να πω ότι αν οι Πολωνοί πιλότοι δεν είχαν πετάξει μαζί με την βασιλική αεροπορία, πολεμική αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καθολικότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Εδώ έχουμε παραβίαση του κοινοτικού και ακτιμένου όταν ε, ε, αναφερόμαστε σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει ενδελεχέστατα να μελετούμε τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, τι περιμένουμε, θα πω εγώ στην Επιτροπή τι περιμένω ε, μετά από μια τέτοια παρουσίαση να θεωρήσω ότι μπορεί να υπάρξει, να ακολουθήσει καριέρα στην πολιτική. Ευχαριστώ τον κύριο Κάσμαν. Δεν μα έχει ακούσει προηγουμένω, αλλά να πούμε ότι όλοι οι συνάδελφοι ζήτησαν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να συνεχιστεί η συζήτηση. Και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρέμβαση του ακριβώς πρόσθεσε ότι ίσως μερικά σημεία και μερικά στοιχεία νέα προκύπτουν από τι σημερινές παρεμβάσει και ίσως καλό θα ήταν να τα προσθέσουμε στην ανακοίνωση που με ιδιαίτερη, ας το πούμε, αγωνία περιμένουμε. Συμφωνούμε με τον συναφέρο Βάλιαν ότι θα πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να εξετάσουμε το θέμα και ότι θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες όλα αυτά τα θέματα που αναπτύχθηκαν και επίσης αποδεχόμενοι και αυτό που ζήτησε ο αναφέρον να δούμε και πάλι τα έγγραφά τους σε αυτή την ε, ιδιαίτερα πλούσια αναφορά του και θα μπορούσα στην Επιτροπή ακριβώς να μπορέσουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ακριβώς για να δούμε μέχρι που φτάνει η αρμοδιότητά μας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γενικά σχετικά με την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους Πολωνίας και Λιθουανίας ε, γιατί μας βοήθησαν και για την παρουσία τους ε, και για τα στοιχεία που μας έδωσαν. Ξέρουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη βοήθειά σας την περαιτέρω για άλλες διευκρινήσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, στην επόμενη αναφορά. Εδώ αλλάζουμε θέμα. Πού πάμε. Στην προστασία της υγείας, ε, την 660 του 2011 της Άννας Σπύρα, παρούσα. Έχει το λόγο για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα σχετικά με την αναφορά της. Ναι. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αφορών. Αυτός είναι ο γιος μου ο Όσκαρ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου προσφέρατε σήμερα τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την αναφορά μου για θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας σχετικά με την κοίηση και τον τοκετό. Είναι η φωνή μιας μητέρας που ακούτε είναι όλοι κορασμένοι, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους γονείς η υγεία των παιδιών τους. Αλλά τα 10% των νεογέννητων, των νεογνών, χρειάζονται βοήθεια και κατά τη διάρκεια ε, της γέννησης και μετά. Και ένα υψηλό ποσοστό ακριβώς 100% ε, δεν ζυγίζει ούτε ένα κιλό και κατηγέννηση ακριβώς. Επίσης υπάρχουν προβλήματα όμως και περισσότερα στις μητέρες και έχουμε πόνους ε, και επηρεάζουν τα πράγματα το ενόπνευμα και ο καπνός. Εδώ χρειάζεται ο γιος μου 24 ώρες το 24ωρο φροντίδες σε ειδικευμένο ε, πρόωρο νεογνών πολωνικό νοσοκομείο γεννήθηκε και δεν ε, δέχτηκε τις απαραίτητες φροντίδες και υπήρξε υπερεμία στον εγκέφαλο ε, και εγκεφαλική παραλυσία κλπ. Εδώ πονάω, πονάω σαν μητέρα να βλέπω την κατάσταση του, του γιού μου να χειροτερεύω και να ρωτιέμαι συνεχώς μετά από το δικό μου το θάνατο ποιος θα ασχοληθεί μαζί του. Και γι' αυτό ακριβώς δίνω μάχη, δίνω μάχη για θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων ε, και στην Πολωνία και στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο έχουμε 500.000 γεννήσεις πρόορες και γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς ε, μια περιγεννητική φροντίδα και να επηρεάσουμε θετικά το 18% της ευρωπαϊκής κοινωνίας. διότι ε, ε, διαφορετικά έχουμε χρόνιες ασθένειες όπως εγκεφαλική παραλυσίες, πολλά προβλήματα, κινητικά κλπ. Και αυτά τα προβλήματα και βαρύνουν και τα παιδιά, αλλά και όλη την οικογένεια, γιατί υπάρχει νευρική εξάντληση και χρόνιες παθήσεις των ε, γονέων και ε, δεν είναι και απαραίτητη υψηλή παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας. Άρα λοιπόν επηρεάζει και υλικά τα πράγματα. Η μητέρα, ας πούμε, δεν μπορεί να δουλέψει και αυξάνεται ο αριθμό των διαζυγίων, δυσκολίες στον ε, οικογενειακό προγραμματισμό γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες ε, που οφείλονται από τα προβλήματα του νεογνού και προβλήματα όπως είπαμε οικονομικά και συνέπειες οικονομικές για το σύνολο της κοινωνίας ε, και μια μείωση γενικά της παραγωγικότητας στη χώρα. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω την κυρία εδώ που είναι από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τα πρόωρα νεογνά η οποία και μετά από μένα θα λάβει το λόγο. Πέρασαν 12 χρόνια από τη γεννήση του παιδιού μου αλλά είναι πάντα ένα τραύμα για μένα εγώ καλούσα το γιατρό γιατί πονούσα, αλλά δεν ερχόταν, δεν ερχόταν ποτέ. Και ευτυχώς υπήρξαν δύο άτομα από δίπλα που με βοήθησαν μέχρι τέλος στη γέννηση του παιδιού μου. Και είδα το παιδί μου ένα κιλό 400 γραμμάρια και μετά δεν ε, ανέπνεε. Εάν είχε τις απαραίτητες φροντίδες, τότε δεν θα είχε υποστεί τις ζημιές ε, μετέπειτα και θα πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά μας το δικό μου. Ε, αλλά ένας ακριβώς από τους γονείς δεν μπορεί να εργάζεται πλέον και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό σαν συνέπεια και μερικές φορές έχουμε και διαζύγια γιατί ε, τα παιδιά, οι μητέρες βρίσκονται μόνες, ε, εγκαταλείπονται να μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους και αυτά φυσικά και πνευματικά επηρεάζει την κατάσταση στις γυναίκες αυτές. Το Επιστημονικό Συμβούλιο υιοθέτησε σωστές συστάσεις για την περιγεννητική φροντίδα, αλλά οι συστάσεις αυτές δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, γιατί δεν υπάρχουν δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις ε, για, την... τον επόμενο χρόνο οι αρμόδιοι για θέματα μευτικής θα προωθήσουν ρυθμίσεις δεσμευτικές και κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να έχει τις απαραίτητες περιγεννητικές φροντίδες κάθε γνώ. Δεν θα πρέπει να εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη περίπτωση, δηλαδή ένα νοσοκομείο ή μια χώρα στην οποία γεννιέται το παιδί αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Πολωνίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με αυτό, γιατί έτσι έχουμε ορισμένα πρότυπα στάνταρτ που να είναι και δεσμευτικά. Και αυτό έχει σημασία για τα μελλοντικά παιδιά που θα γεννηθούν χάρη σε αυτή την περιγεννητική φροντίδα στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να έχουμε μια υψηλή ποιότητα φροντίδα για να μπορούν να έρχονται στον κόσμο υγιή και κάθε οικογένεια να χαίρεται την ανάπτυξη του παιδιού της που να είναι υγιές. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να υποστηρίξετε την έκθεσή μου, την αναφορά μου. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα κάπως, αλλά επίσης και η κυρία εδώ δίπλα μου, μήπως θα μπορούσε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρετε τώρα το λόγο. Πολύ ωραία. Sicherheitshalber spreche ich in meiner Sprache, θα προτιμήσω στη γλώσσα μου να μιλήσω υποστηρίξω ενεργά την κυρία Σπάιντερ από την αρχή του αγώνα της και εγώ είχα τέτοιο ατύχημα και είμαι ηγετικό τέλο το 2008 του Ιδρύματος για την Περιγενική Βοήθεια και τη Βοήθεια στον Τοκετό και προσπαθούμε να κάνουμε συστάσεις. Χρειαζόμαστε κάθε στήριξη ούτως ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά στην Ευρώπη. Η κατάσταση είναι ότι 5 εκατομμύρια παιδιά γεννούνται κάθε χρόνο, 2 εκατομμύρια Επιπλέον, ε, δεν γεννιούνται ζωντανά. 25.000 παιδιά γεννιούνται νεκρά και 90.000 έχουν μεγάλα προβλήματα και 500 παιδιά γεννιούνται κάθε μέρα ε, πριν το τέλος ε, της εγκυμοσύνης Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε συγκεκριμένες χώρε και τα ποσοστά μπορεί να μοιάζουν διαφορετικά γιατί δεν έχουμε το σωστό σύστημα εγγραφή σε Μητρώα. δεν ε, εγγράφονται σωστά ε, στα Μητρώα τα παιδιά. Κάθε εβδομάδα από την 37η και μετά έχει σημασία πόσο θα κρατήσει η εγκυμοσύνη μετά την 37η ε, εβδομάδα για το αν θα μπορέσει να επιζήσει, δηλαδή κάτω το κετό για το αν θα έχει προβλήματα αναπηρίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει περιγυνητική βοήθεια πολύ ψηλού επίπεδου και αυτή η περιγυνητική φροντίδα να γίνεται από υψηλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό γιατί στη τελευταία ανάλυση έχουμε μόνο έναν εγκέφαλο, έχουμε μόνο δύο πνεύμονες, μία καρδιά. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναπτυχθούν αρκετά αυτά τα όργανα και να βοηθηθούν για να γίνει υγεία στο παιδί. Η υγεία βεβαίως έχει να κάνει και με τη φροντίδα ε, μετά τη γέννηση. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση στη χώρα σας. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία και την Αυστρία είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, ενώ οι βόρειες χώρες έχουν πολύ καλύτερη φροντίδα και πολύ περισσότερη ενημέρωση και έχουν υψηλό επίπεδο γενικά φροντίδας, τα οποία εφαρμόζονται σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για την ε, γέννηση προώρων και γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν ομάδα πίεσης είναι δυστυχώς ε, το κάπνισμα, η κατανάλωση ινοβηματοδών, τα ναρκωτικά. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Ε, μετά έχουμε διάφορες μολύνσεις, όχι επαρκή φροντίδα και κυρίως όχι επαρκή πληροφόρηση των εγγύων. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο ενημέρωσης ε, των εγγύων τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολλές επιπλοκές και πολλές φορές κατά τη γέννηση υπάρχει έλλειψη ε, οξυγόνου. Αυτό προκαλεί βαριές ε, διανοητικές αναπηρίες μέχρι και εγκεφαλική παραλυσία. Αυτό δημιουργεί δυσχέρες μετά για την εκπαίδευση των παιδιών και χρονικές ασθένειες, για παράδειγμα δεν έχουν οριμάσει αρκετά η καρδιά και οι πνεύμονες Έχουμε κατόπιν ε, χρόνιες ασθένειες και έχουμε μελέτες που αποδεικνύουν ότι 10% των προώρων έχουν, διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο να ε, πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Ο εγκέφαλος ε, αναπτύσσεται ακριβώς την περίοδο που γεννιούνται τα πρόωρα. Οπότε, εάν υπάρξει ε, ένταση και στρες κατά τον δοκετό, κατά τον δοκετό τότε έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν ότι αν δεν υπάρξει καλύτερη φροντίδα και δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι 500.000 πρόωρα γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και δεν έχουν όλα βέβαια βαριές αναπηρίες Αλλά πρέπει να καταπολεμήσουμε το γεγονός αυτό και να δώσουμε στο 10% των παιδιών αυτών ε, μια καλύτερη δυνατότητα επιβίωση και ποιότητα ζωή. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε μια ανατολική χώρα που δεν υπάρχουν ε, επαρκείς συνθήκε και εξοπλισμό. Ε, χορηγείται οξυγόνο, αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς ε, οθόνες που να ενημερώνουν για το πώς δίνεται το οξυγόνο γιατί αν δώσουμε υπερβολικό οξυγόνο μπορεί να οδηγηθεί το παιδί σε τυφλότητα και εκεί σε αναπηρίες. Σε... Και κατόπιν βέβαια ε, ε, υπάρχουν δυσχέρειες και στις σχέσεις με τους γονείς. Έχουμε κατόπιν λοιπόν πολλές ασθένειες τα παιδιά που έχουν διάφορε αναπηρίε. Α, και πάλι μιλάω πολύ γρήγορα. Α, καλά. Έχουμε λοιπόν διάφορε αναπηρίε που ε, δημιουργούν μακροπρόθεσμο κόστος, αλλά ακόμη και ελαφρές αναπηρίες που μπορούν να έχουν κάποια προώρα, φυσικά μειώνουν την εκπαίδευσή τους και την ε, απόκτηση προσόντων για την επαγγελματική του ζωή, καθώς και για κοινωνικές, και κοινωνικές επιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορες μελέτες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μια μελέτη κατέδειξε ότι μπορεί να μειωθεί κατά πολύ το κόστος εάν ένα προώρο γεννηθεί μια εβδομάδα αργότερα. Κάθε μέρα μετράει. Εδώ έχουμε μια αμερικανική μελέτη όπου αποδεικνύεται ότι δεν ε, μας ενδιαφέρει μόνο το άμεσο κόστος αλλά και το μακροπρόθεσμο κόστος. Για παράδειγμα, έχουμε επανεισαγωγές στο νοσοκομεία για διάφορους λόγους. Τετραπλασιάζεται έτσι το κόστος. Κάθε πίνακας δείχνει τι τεράστιο συμπληρωματικό κόστος δημιουργείται από τα πρόωρα. Όσο αργότερα γεννηθούν τα πρόωρα, τόσο καλύτερα. Αλλά και η οικογένεια και η κοινωνία επιβαρύνονται ιδιαίτερα το ακούσατε ήδη. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να εργαστούν. Υπάρχει ψηλότερο κίνδυνο ε, διαζυγίου στι οικογένειε αυτές. Οι οικογένειε αυτέ δεν κάνουν κατόπιν ε, περαιτέρω παιδιά. Υπάρχει λοιπόν τρομερή απώλεια για την ε, ευρωπαϊκή, κοινωνία του μέλλοντο. Μακροπρόθεσμα λοιπόν για την κοινωνία, αν ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία κόστου. καταλαβαίνετε πώ έχουν τα πράγματα. Ευρωπαϊκά πρότυπα Δεν είναι μόνο δική μας υποχρέωση. Υπάρχει πολύ ψηλό κίνδυνος και για τους μετανάστες. Οι μετανάστες ε, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να, κάνουν, να γεννήσουν προώρα γιατί και λόγω γλώσσας είναι δυσκολότερο να τους υποστηρίξουμε, να τους ενημερώσουμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά από ποια κουλτούρα προερχόμαστε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Να ορίστε μια φωτογραφία του γιού μου. Γεννήθηκε 550 γραμμάρια. Είναι 15 ετών τώρα. Αυτό το δεντρίλιο που βλέπετε πίσω από την οικογενειακή ε, φωτογραφία είναι δεντράκι που ε, ε, φυτέψαμε πάνω στον τάφο της κόρης μου η οποία θα έχει γεννηθεί αν είχαμε αυτά τα πρότυπα θα έχει επιζήσει δηλαδή πιστεύουμε λοιπόν ότι στο μέλλον πρέπει να παλέψουμε για υγιή παιδιά και υγιείς γεννήσεις ευχαριστώ σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Γκέβελ παρακαλώ παρακαλώ σύντομα η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εντάξει. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχάς ευχαριστώ τις ομιλήτρες γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση όπως την παρουσίασαν. Η Κομισιόν όμως ε, έχει πολύ περιορισμένες ε, δυνατότητες των τομέα της υγείας μπορεί να δώσει πληροφόρηση και το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Και συνεργάζεται με διάφορα προγράμματα σε μεγάλο βαθμό. Τα προγράμματα αυτά και οι πληροφορίες είναι στη διάθεση και των κρατών μελών. Αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να διαδώσουν αυτή την πληροφόρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επιδράσει από αυτού καθόλου. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την περαιτέρω διάθεση και χρήση αυτής της πληροφόρησης. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, αναγνώριση των προσπαθειών της των δύο κυριών για τη μάχη που δίδουν εδώ και χρόνια για ευρωπαϊκά πρότυπα ακριβώς σχετικά με την κοίηση και τα νεογνά. Εδώ θεωρώ ότι αποτελεί χρέος κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους για παρόμοια πρότυπα. Παρακαλώ την κυρία Σπύρα να μου πει τα εξής. Αρκετές φορές λένε ότι η υιοθέτηση παρομοίων προτύπων συνεπάγεται κόστος, υψηλό κόστος. Αλλά επίσης αναφέρεται ότι τελικά μακροπρόθεσμα έχουμε μία μίσο του κόστους. Τι λέτε σχετικά με αυτό. Ε, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η σημερινή αναφορά της κυρίας Πύρα αφορά μια ρύθμιση ευρωπαϊκή για την περιγενική φροντίδα και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχω επαφή με την κυρία Σπύρα και βλέπω τι ακριβώς κάνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η αναφορά της κυρίας Σπύρα, όπως επίσης και το πρόβλημα αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί βλέπουμε ότι δεν υπήρξαν ρυθμίσεις και δεν ε, υπήρξαν φροντίδες από σμένα κρατημέλη για την δημιουργία παρομοίων προτύπων. Είναι φροντίδες ιατρικές ε, άμεσης ε, κατάλληλης εφαρμογής από πλευράς νοσοκομείων και δεν δίδονται οι φροντίδες όπως πρέπει κατά τη διάρκεια της γέννησης των νεογνών ακριβώς αυτά τα κενά τα νομικά οδήγησαν σε αυτά τα προβλήματα. Δύσκολο τώρα είναι να πει κανείς ε, αν αυτό που κάνει το ιατρικό, το ιατρικό προσωπικό είναι και η κατάλληλη ενέργεια για, για τις ε, καλύτερες συνθήκες ε, για τα νεογνά. Εδώ Αυτά που λέει η κυρία Σπύρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τις φροντίδες αυτές για τα νεογνά, κυρίως για τα πρόωρα. Εγώ υποστηρίζω την αναφορά και την προσπάθεια της κυρίας Πύρα και το αίτημά της ώστε επιτέλους να υπάρξουν κοινοτικά πρότυπα στην Ευρώπη ε, για την διάρκεια της και για τη γέννηση. Και θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι την κυρία Σπύρα. Σε ποιο, σε τι πλαίσιο θα πρέπει να εισαχθούν αυτά τα καινούργια πρότυπα, τι μορφή θα πρέπει να έχουν και τι θα αλλάξουν αυτά τα πρότυπα. Και ακόμα κάτι, εάν όλα αυτά ίσχυαν ήδη, ίσως ο γιος σας θα είχε περισσότερες πιθανότητες να ζει κανονικά όπως και τα υπόλοιπα παιδιά και η κυρία Μάντερ από δίπλα. Σας θα ήθελα να ρωτήσω το εξής εκείνη. Εσείς ε, πώς σκέφτεστε, τι μορφή θα πρέπει να έχουν αυτά τα πρότυπα για την περιγεννητική φροντίδα των νεογνών και δυστυχώς κάποιος κάποιο συνάδελφο που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα εδώ. Ακριβώς τι δυνατότητες υπάρχουν να μεταβληθούν αυτά τα πρότυπα για τις προγεννητικές και μετηγενετικές φροντίδες. Και τα πρότυπα αυτά τι συνεπάγονται, ιδιαίτερα υψηλό κόστος, υψηλότερο κόστος για το σύστημα το υγειονομικό. Ναι, το λόγο έχει η κυρία Σπύρα για να απαντήσει, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Ε, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, έστω και αν υπευλήθησαν αρκετά ερωτήματα. Η εισαγωγή ε, προτύπων ε, και νομικών ε, υποχρεώσεων ή δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά την περιγενετική περίθαλψη. Νομίζω ότι ε, θα ε, μείωναν την ε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε λόγω του ελλειπούς εξοπλισμού. Τώρα θα συμφωνήσουν και οι πιο φτωχές χώρες γι' αυτό, γιατί εδώ μιλάμε και για εξοπλισμό ε, στα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν όμως να επιτρέψουμε 10% των πρόωρων ε, παιδιών που, ζητού, που απαιτούν μάλλον ε, συνομιλική πρόσβαση οξυγόνου ή θερμοκοιτίδες να μην έχουν την δυνατότητα να επιζήσουν κανονικά, να, να καταδικάσουμε τα παιδιά αυτά να ζουν όπως ζει ο γιος μου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει κάθε μευτική μονάδα ε, τον εξοπλισμό το βασικό, δηλαδή η θερμοκοιτίδα και ε, δυνατότητα ε, παροχής οξυγόνου. Υπάρχουν καταστάσεις όπου οι γυναίκες δεν ξέρουν πού να αποτανθούν δεν ξέρουν αν ε, σε κάποιο νοσοκομείο υπάρχει θερμοκριτίδα και αν αυτή η θερμοκριτίδα θα είναι διαθέσιμη, αν γνωρίζουν ότι η κοίησή τους θα ολοκληρωθεί πρόωρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάχα συστάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συστάσεις ε, που αφορούν και τη συμπεριφορά ε, του ιατρικού προσωπικού, αλλά όχι τον εξοπλισμό. Αυτό αφήνεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως και ο εξοπλισμός είναι θεμελιώδους σημασίας. Οι γονείς, ε, όπως εγώ η ίδια, ε, ε, πρέπει τελικά να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να αναλάβουν, να αντέξουν αυτό το βάρος διαζύγια. Τα διαζύγια είναι πολύ περισσότερα σε αυτές τις ε, περιπτώσεις και τελικά ποιος πληρώνει το κόστος. Θα πρέπει ακόμα και χρηματοδοτικά να βοηθηθούν αυτοί οι ευάλωτοι γονείς γιατί διαφορετικά ε, θα μειωθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό των γεννήσεων στην Ευρώπη. Οι γονείς ε, δεν θα θέλουν μπροστά στην αβεβαιότητα αυτή να γεννήσουν παιδιά. Θα πρέπει η περιγεννητική περίθαλψη να είναι ικανοποιητική. Δεν αναφέρομαι σε όλες τις διαδικασίες και σε όλες τις μορφές περίθαλψης. Ενδεχομένως η στήριξη τουλάχιστον της ε, ε γυναίκας. Αυτή είναι ε, η οποία αποφασίζει για το μέλλον του παιδιού της. Ε, σαν μητέρες εμείς κάνουμε πολλά, αλλά μερικές φορές δεν καταφέρνουμε ούτε να φτάσουμε μέχρι το νοσοκομείο μέχρι την ε, κλινική. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα. Μερικές φορές δεν έχουμε το χρόνο ούτε καν να φτάσουμε μέχρι το μεευτήριο. Δεν είναι εύκολο να απαντήσω βέβαια σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι απαντήσατε στα κυριότερα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν και εν πάση περιπτώσει ε, και όλα τα σχετικά με αυτό το με αυτή την αναφορά ζητήματα μας οθούν στο να την κρατήσουμε ανοιχτή. Θα ζητήσουμε ε, και μια ειδική αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοώντας βεβαίως τα όρια της θεσμικής δικαιοδοσίας ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια πρωτοβουλία απέναντι στις τοπικές αρχές και ταυτόχρονα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο όλες, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αφορούν το ζήτημα αυτό. Πολλές είναι οι δυνατότητες υποβολής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ας πούμε, για την προώθηση του δικαιώματος στην υγεία και αυτό δίνει την δυνατότητα και στην Κομισιόν να έχει μια πιο αποφασιστική παρέμβαση απέναντι στις χώρες αυτές οι οποίες δεν καταφέρνουν να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ε, και που έρχονται εδώ με ιδιαίτερα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία χωρίς να αντιμετωπίσουμε μόνο συγκινησιακά ε, τα ζητήματα τα οποία θίγουν οι δύο αναφορές. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό το ζήτημα, να εξακολουθήσουμε από κοντά, να παρακολουθούμε τις ε, αναφορές αυτές. Εάν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν θα ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή μας συζήτηση για αυτές τις δύο αναφορές. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τις ε, ε, την κυρία Σπύρα και την εκπρόσωπο της της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ε, για τα πρόωρα παιδιά και ολοκληρώνουμε την συζήτηση της αναφοράς. Έχουμε τώρα την γνωμοδότηση της κυρίας Βάλεαν, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε μας ζητήθηκε να γνωμοδοτήσουμε ε, για το ε, πρόγραμμα 14-20 ε, από την αρμόδια καθήλια επιτροπή που είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ε, πολλές αναφορές ε, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες στην προσπάθειά τους για ελεύθερη κυκλοφορία. Αφορά αυτό το ζήτημα 25% περίπου των παραδεκτών αναφορών. Το 2010 εκπονήθηκε έκθεση σχετικά με την αποτελεσματική πορεία της Ευρώπης προς την πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, ε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, καθυστερήσεις στις διοικητικές ε, διαδικασίες, στην έκδοση καταγραφής σε μια άλλη χώρα, η δυσκολία στην έκδοση ταυτοτήτων κτλ. Αλλά επίσης και όσον αφορά την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Την τελευταία χρονιά είχαμε 63 διαδικασίες επί παραβάση ε, για θέματα σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών που διαβιούν σε άλλη χώρα. Ε, σε μεγάλο ποσοστό τους ε, οι πολίτες ε, δηλώνουν ότι, δεν έχουν, ότι έχουν ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η ελλειπής πληροφόρηση λοιπόν αποτελεί μία, αν όχι την, κυριότε, το κυριότερο εμπόδιο, το κυριότερο πρόσκομα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πληροφόρηση λοιπόν και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Διαρκής παρεξήγηση για τα ζητήματα αυτά υπάρχει σχετικά με το ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή τη, αν μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι, αν εμπίπτει στι αρμοδιότητε στο πεδίο εφαρμογή ή όχι. Είναι γεγονός πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ε, ε, διακρίσεις όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, ε, η οχι αν εμπιπτει στι στο πεδιο εφαρμογη η οχι ειναι γεγονος παντως οτι εξακολουθουν να υπαρχουν σημαντικες διακρισεις οσον αφορα τους ευρωπαιους πολιτες επισης η αντιμετωπιση των γυναικών είναι ιδιαίτερα προβληματική τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν ακόμα να χαίρουν πλήρους ισότητας παρά ε, των περιαντιθέτου αναφερομένων στη, στη, στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, όσον αφορά τώρα τα δικαιώματα ε, των εγκατάστασης και το δικαίωμα του επιχειρήν, στην προκείμενη περίπτωση έχουν έχουν υπάρξει πάρα πολλά προβλήματα, ε, τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν μονάχα με την σωστή κατάρτιση και τα, τη δημιουργία ε, διασυνοριακών και διεθνικών προγραμμάτων συνεργασίας και δικτύων. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν έρευνες οι οποίες θα αποτελέσουν βάση ε, για την περαιτέρω συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πρόγραμμα 2014-2020 ε, διαδέχεται τρεις προηγούμενες προσπάθειες που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, την μείωση των, της διακριτικής μεταχείρισης των μειονοτήτων και την ισότητα των φύλων που έχουν οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και με την βοήθεια και του προγράμματος Progress μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη και πιο ευέλικτη χρήση των ε, χρηματοδοτικών εργαλείων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και απλούστευση των διαδικασιών και εναρμόνιση των κανόνων. Το πρόγραμμα αυτό θα ε, αποσκοπεί και στην καλύτερη ε, κατανομή των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα στα πλαίσια πλαίσια καλύτερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού. Ε, υπάρχουν κάποιοι ετούντες καθώς επίσης μεμονωμένοι αλλά και κάποιες οργανώσεις οι οποίες ε, αναφέρονται στη δυσκολία πρόσβασης ε, στα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως όταν πρόκειται για μικρές εταιρείε ή μικρές μικροβιενετικές οργανώσεις. Χρειάζεται και διασυνοριακή κατανομή των χρηματοδοτήσεων όχι μονάχα σε μεγάλες και διευρωπαϊκές οργανώσεις αλλά και σε μικρότερες οργανώσεις. Ο 8 Μαΐου είναι η προθεσμία για την γνωμοδότηση, ή ε, συγγνώμη, για την έκθεση στην αρμόδια καθήλια επιτροπή και στην, ε, στην Ολομέλεια του Ιουλίου θα έρθει το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι Βαλεάν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ε, θέμα αυτό. Ε, πιστεύω ότι στην επόμενη ε, συνεδρίαση θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο και εντωμεταξύ όμως ε, θα έχετε οπωσδήποτε ε, και κάποια επιπλέον στοιχεία, θα έχετε συμβολές και από τους συναδέλφους. Άλλωστε και η σημερινή συζήτηση συνέβαλε στο να κατανοήσετε πώς προς η κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε. Έχουμε τώρα την ε, έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο. Θα δώσω τον λόγο στον ε, κύριο Μπουλάν ε, που ήταν επικεφαλή τη διερευνητική αυτή επιτροπή. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. η συνάδελφο, κανονικά θα λάμβανε το λόγο για αυτό το θέμα, αλλά εντάξει να σας κάνω μια περίληψη τι ακριβώς μέχρι τώρα σημειώσαμε σαν κύριο σημείο, τα πρακτικά δηλαδή μια αποστολής, μιας επίσκεψης με την κυρία Λιώτοβα και στην ομάδα που επισκέφθηκε το Βερολίνο και ήταν ε, το βασικό κείμενο βάσης εργασίας και θα επιτρέψει στα μέλη τη αντιπροσωπείας να μπορέσει τελικά να το τροποποιήσει αυτό το κείμενο για να υποβληθεί να επιτευχθεί στην Επιτροπή Αναφορών μια συνένεση για την έκθεση αυτή και μετά να παρουσιαστεί εδώ και να ψηφιστεί και μετά ακριβώς το κείμενο να μπορέσει να γίνει δημόσιες ε, παρουσία, να γίνει γνωστό για την εργασία εδώ και για την αντιπροσωπεία η οποία μετέβει στο Βερολίνο. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Ίσως θα μπορούσαμε σήμερα στο παρουσιάσουμε αυτό το κείμενο, αλλά δεν είχαμε και το χρόνο να εργαστούμε αποτελεσματικά. Πάντως συμφωνήσαμε όσον αφορά τη μεθοδολογία και το μόνο που μας μένει εδώ στην ε, ε, ομάδα αυτή εργασίας να επιφέρουμε τις απαραίτητες μετατροπές και είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Ε, δεν περίμενα να πάρω το λόγο τόσο σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Φιλίπ Μπουλάν για την παρουσίαση του περιεχομένου. Αυτή την οδό πρέπει να ακολουθήσουμε να έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε οι μεν τις ε, θέσεις των δε και να τις ε, προσεγγίσουμε. Ο Φιλίπ ε, τα είπε πολύ σωστά και το χρονοδιάγραμμα μας επιτρέπει πιστεύω να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Γεια. Σύντομα. Ευχαριστώ τον Φιλίπ Μπουλό σωστή η διαδικασία που προτείνει. Μια παράκληση. Στην επόμενη συνεδρίαση να έχει υποβληθεί η έκθεση από την ομάδα εργασίας. Ομοφωνία είναι πάντα ο καλύτερος ε, τρόπος. Αναμένουμε λοιπόν, προσβλέπουμε στο κείμενο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα εργασίας ε, εγκαίρως θα μας το υποβάλει. Ε, νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να γίνει σχετικά σύντομα. Λεγκούτο. Σύντομα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μας έχει υποβληθεί. Ε, θα έπρεπε να κλείσει όσο δυνατόν πιο σύντομα. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές λογικές ε, συστάσεις ε, στο έγγραφο εργασίας. Αλλά έχουμε χρονοτριβήσει υπερβολικά. Νομίζω ότι επήγει. Μποστινάρου. Μια πρόταση. Χαιρετίζω αυτήν την ε, σόφρονα άποψη. Να κάτσουμε μαζί. Να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που να είναι επωφελής για την Επιτροπή μας και την αξιοπιστία της εργασίας, μου. της εργασίας μας. Χαίρομαι λοιπόν για αυτό το αποτέλεσμα. και θα πρέπει να είναι παράδειγμα και για το μέλλον αυτή η διαδικασία να αποφύγουμε συγκρούσεις στο μέλλον. Η Πρόεδρος, συνοψίζοντας τα όσα είπατε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφε δεν είναι εδώ η κυρία Γιώτοβα. Από ό,τι κατάλαβα είναι, θα συμφωνήσετε, α, λεπτό, ήρθε Δύο-τρία λεπτά ακόμα, κυρία Γιώτοβα, έχουμε στη διάθεσή μας πριν να ολοκληρωθεί η συνάντησή μας. Αν θέλετε, έχετε το λόγο. Уважаеми колеги, днес ще ви информирам за хода на работата по документа от Не, θα, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια σχετικά με την εργασία που κάναμε στην ε, διερευνητική αποστολή στο Βερολίνο σχετικά με τους ε, μικτούς γάμους. Ε, ακόμα και όταν πρόκειται για ανθρώπους ίδιας εθνικότητας βλέπουμε ότι υπάρχει κλιμάκωση των ε, αντιδράσεων όσον αφορά την κυδαιμονία των παιδιών Υπάρχουν ε, περιπτώσεις βεβαίως όπου οι γονείς έχουν πλήρη άγνοια του νομικού συστήματος ε, και των νομικών ε, αρχών. Υπάρχει σημαντικός αριθμός αναφορών στις περισσότερες από αυτές ε, αναφέρεται ότι ο τρόπος ε, αντιμετώπισης ε, είναι διακριτικός και καταχρηστικός. Ήδη από το 2007 έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα. Αυτά μάλλον όχι οι αναφορές οι οποίες σχετίζονται με το θέμα αυτό απέναντι σε γονείς δηλαδή που δεν είναι Γερμανοί και των οποίων τα παιδιά δεν μπορούν μπορούν να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Ε, ήρθαμε σε επαφή με ε, εκπροσώπους ε, των, του Δικαστηρίου των Ανηλίκων. Ήρθαμε σε επαφή και με εκπροσώπους του Φορέα για την Νεολαία και ε, ε, γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε ακόμα προετοιμάσει το έγγραφό μας. Ε, έπρεπε να δουλέψουμε πολύ, συναντηθήκαμε πολλές φορές και μεταξύ μας. Έχουμε, οργανώ... έχουμε ήδη εκπονήσει ένα προσχέδιο του εγγράφου, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι ευαίσθητο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε βεβαίως και στην... στα εσωτερικά της γερμανικής νομοθεσίας ή να μην σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Από την άλλη στην πλευρά βεβαίω θέλουμε να βοηθήσουμε τους ε, αναφέροντες που ζητούν βοήθεια από εμά. Πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούμε να λαμβάνουμε επιστολές από πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα με τις ε, υπηρεσίες νεολαίας στην Γερμανία προσπαθούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό ε, και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε σε συνενετική βάση ένα κείμενο το οποίο θα σας υποβάλουμε ως ονούπο. Ε, Άρα λοιπόν, για τη συνάντησή μας ε, την επόμενη θα εντάξουμε στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του κειμένου. Πίλαντ. πολύ σύντομα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπήρξε κάποια κινητικότητα για το θέμα αυτό. Τρία πράγματα με ενδιαφέρουν. Πρώτον, η αναφορά θεωρήθηκε παραδεχτή όσον αφορά το περιεχόμενό της, διότι ε, έχει ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη διαδικασία που καταγγέλλεται να θίγονται πολίτες της Ένωσης. Δεύτερον, ότι ήταν λίγος ο χρόνος στην Αλφεγιάρ. Έκανε ό,τι μπορούσα. Επανειλημμένα είπαμε. Χρειαζόμασταν δύο μέρες. Αλλά η Επιτροπή θέλησε να πάμε μόνο μία μέρα. Δεν ήταν επαρκής ο χρόνος. Μπορέσαμε λοιπόν ε, πολύ λίγο να μιλήσουμε με τους θυγωμένους. Και τρίτον, Έχω πάει σε αρκετές αποστολές για εξέβρεση στοιχείων, fact-finding. Είναι τα μάτια και τα αυτιά τη Επιτροπής μας επιτόπου σε κάποιο θέμα. Και αυτά που βλέπουμε μετά είναι αντικείμενο της έκθεσης. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψετε, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, για τα πορίσματα της έκθεσης να υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροπολογιών να ψηφίσει συνολικά η Επιτροπή. Στείλαμε εκπροσώπους, αλλά η συνολική αντιμετώπιση του θέματος είναι υποχρέωση της συνολικής Επιτροπής. Η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βίλαντ. Αυτή είναι η άποψή του. Ήταν μέλος αντιπροσωπείας και η άποψή του δεν δεσμεύει τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας. Αυτό το έγγραφο που θεωρήσαμε σαν έγγραφο εργασίας ψηφίστηκε απέναντι σε ένα άλλο πολύ πιο περιληπτικό κείμενο. Και το κείμενο αυτό εργασίας, ε, το οποίο συμφώνησαν τα περισσότερα μέλη της αντιπροσωπείας ακριβώς, γιατί είχε τις περισσότερες προτάσεις των μελών, τα οποία μετέβησαν στο Βερολίνο. Πρώτο σημείο. Να πάμε στο δεύτερο για μια ψηφοφορία για να είναι τα πράγματα όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και δημοκρατικά ανάμεσα σε εκείνου που εργάστηκαν για το έγγραφο αυτό και τρίτο σημείο και εδώ δεν συμφωνώ και απόλυτα με αυτό που ο κύριος Βίλαντ ε, προτείνει. Ποιες είναι οι συνήθειες σχετικά δεν γνωρίζω. Αλλά στην ομάδα αυτή εργασίας Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συνένωση μέσω δικών μας εσωτερικών αυτής της ομάδας τροπολογιών. Και έτσι, όταν το οριστικό κείμενο, αποτέλεσμα της συνένεση συμβαστικών λύσεων κλπ. υποβληθεί στην ε, Επιτροπή Αναφορών, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ψηφίσει κανονικά υπέρ κατά αυτή η Επιτροπή. Αλλά ε, πώς μέλη τα οποία δεν εργάστηκαν πάνω σε αυτά, δεν είδαν, δεν ε, τα μελέτησαν όλα αυτά διαδοχικά, τα διάφορα που προέκυψαν. Εντάξει, γιατί ο καθένας σας ασχολήθηκε και με άλλα θέματα. Λοιπόν, πώς τα μέλη αυτά θα μπορούσαν να τροποποιήσουν αυτό το κείμενο. Και αυτό χωρίς να ξέρουν, χωρίς να ήταν εκεί αυτοί οι μάρτυρες και να είδαν με τα ματάκια τους το τι συμβαίνει. Εντάξει, με κάθε σεβασμό σας τα λέω αυτά, εντάξει, για την Επιτροπή σας αναφορών ε, για ένα κείμενο από την ομάδα εργασίας θα πρέπει να συνταχθεί με μία συνένεση και το κείμενο αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί. Όχι όμως να τροποποιηθεί γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν λογικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, έληξε ο χρόνος, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά, έτσι.